να καλωσορίσουμε την ύπατη εκπρόσωπο Βαρόνι Άστον. Η παρουσία της εδώ είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και ενδιαφέρουσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Διαπιστώσαμε την δυσκολία να φτάσουμε σε κοινή θέση ε, μεταξύ των 27 κρατών μελών, μια θέση που να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική, συνεκτική, αλλά και πιστή στις αξίες και τις αρχές αρχές επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρόνι Άστον, το Σάββατο εσεί συμμετείχατε στη συνάντηση των Παρισίων που προώθησε ο πρόεδρος Σαρκοζή και χθε έγινε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων πολύ πυκνή, με πολύ σημαντικά θέματα και πολύ λεπτά θέματα. Η παρουσία σας σήμερα εδώ λοιπόν είναι ε, άκρος επίκαιρη και μαρτυρά τον διάλογο που θελήσατε να θεσπίσετε με την Επιτροπή μας και μέσω του Επιτρόπου Φίλε και του Γενικού Γραμματέα Βημό. Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι πολλά. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι το πιο σημαντικό και πρώτο. Η... Εξελίξει στη Βοσνία Ζεγοβίνη, έναρξη διαλόγου ανάμεσα στους Σέρβους και τους Κοσοβάρους, η στρατηγική στο Σαχέλ, η κατάσταση στη Σομαλία, αλλά και η φυσική και η πυρηνική καταστροφή που έπληξε την Ιαπωνία. Δεν θέλω να χάσω παραπάνω χρόνο, γι' αυτό σας δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγησή σας. Ε, συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθούμε και να σκεφτούμε τα όσα έχουν γίνει από την τελευταία μας συνάντηση εδώ σε αυτή την Επιτροπή τον Οκτώβριο. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε νομίζω πως οι ρυθμοί των αλλαγών ήταν αδυσόπιτοι. Στη, σε 28 διαφορετικές αποστολές συμμετείχα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτοτε και αυτή τη στιγμή ε, εστιασμός μας ε, σωστά είναι στη Λιβύη τα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλαγές στην νότια γειτονία μας. Ε, όλα αυτά φυσικά επισκιάζουν ό,τι άλλο συμβαίνει και είναι κατανοητό αυτό, αλλά ανέκαθεν ναι, έλεγα πως η γειτονιά μας είναι μια δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πώ ανταποκριθούμε δηλαδή στα γεγονότα στην ίδια μας τη γειτονιά καθορίζει την αποτελεσματικότητα τη Ένωση και φυσικά της νέας υπηρεσίας. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω πως οι σκέψεις μας τελευταίες μέρες ε, βρίσκονται κοντά στον Ιαπωνικό λαό. Είχα μια συνάντηση στο Παρίσι με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα ε, και του εξέφρασα τις ευχές του Κοινοβουλίου και όλων των λαών της Ευρώπης καθώς η Ιαπωνία πρέπει να αντιμετωπίσει τα, τον αντίκτυπο του σεισμού και του τσουνάμι. Όταν ανατρέξουμε στα όσα έγιναν από τον Οκτώβριο, θυμάμαι ότι τα Χριστούγεννα ε, ασχολούμασταν και ανησυχούσαμε πολύ με την ακτή του Ελεφαντοστού. Γιατί είναι μια χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναταραχή και ακόμα δεν υπάρχει επίλυση της κατάστασης ώστε να μπορέσει ο πρόεδρος Βατάρα να αποκτήσει τον έλεγχο της χώρας του. Επίσης συζητούσαμε τη Λευκορωσία και τις ανησυχίες μας για την αξιοπιστία των εκλογών εκεί και κατά συνέπεια την πίεση που ασκήσαμε, τις δύσκολες συναντήσεις που είχαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών Ματινόφ και την εργασία που εξακολουθούμε να κάνουμε ώστε να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης ενώ εξασφαλίζουμε ότι έχουμε επαφές με τον λαό της Λευκορωσίας. Έκτοτε φυσικά Έχουμε εμπλακεί στην ειρηνευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή. Δύο φορέ έχω επισκεφθεί το Ισραήλ, έχω ε, έρθει σε επαφή με τις, ε, την Παλαιστινιακή Αρχή, είχαμε τι συνεδριάσει στο Μόναχο, την ε, συνάντηση των επεσταλμένων εδώ αλλά και οι απεσταλμένοι μας εκεί με επικεφαλή τον ε, Χέλμουτ Σμιτ εδώ συνάντησαν τις αντιπροσωπείες δύο φορές. Δύο φορές συμμετείχα σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την ε, πυρηνική τα πυρηνικά όπλα, προσπαθούσα να προχωρήσουμε όσο γινόταν με τις προτάσεις που υποβάλαμε εμείς, να πείσουμε το Ιράν να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα, να αναγνωρίσει την πολιτική πυρηνική ενέργεια μόνο και ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί τους. Θα πρέπει να σας πω ότι ενώ οι προτάσεις μας εξακολουθούν να συζητώνται και εξακολουθούν να στέλνουν μηνύματα προς το Ιράν, περιμένουμε την απάντησή τους μέχρι σήμερα. Επίσης, ε, ασχοληθήκαμε με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ένα σημαντικό στοιχείο Πολύ περισσότερο τη σήμερα ημέρα. Χθε συνομιλούσα με τον Γενικό Γραμματέα Ράσμου, με τον οποίο έχω τακτικέ επαφέ για να δούμε πώ καλύτερα θα μπορέσουμε να δράσουμε από κοινού. Και επίση ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με το οποίο ασχολούμαι τελευταία, είναι η Μολδαβία και η Περνιστερία. Συζητούμε με τη Μόσχα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις. Από όσο γνωρίζω, πολλοί ε, βουλευτέ παρακολουθούν πολύ στενά την έναρξη των διαπραγματευσεων σερβιας Σερβία-Κωσυφοπεδίου. Πρώτη συνάντηση ήδη έχει γίνει, δεύτερη θα γίνει αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Επίσης φυσικά γνωρίζω ότι ενώ σκεφτόμαστε όλα αυτά τα διαφορετικά θέματα, εξακολουθούμε να οικοδομούμε μια νέα υπηρεσία. Και πιστεύω και νομίζω ότι μπορούμε να αποδείξουμε πλέον ότι στην καρδιά των όσων κάνουμε βρίσκεται αυτή η ιδέα ότι Βρισκόμαστε εδώ για να επιλύσουμε τις διαφορές, να στηρίξουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία, να στηρίξουμε την επιθυμία των λαών, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους και να χαίρουν των διαφόρων ε, ελευθεριών. Γι' αυτό είναι το σημαντικός ο διάλογος μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας, γι' αυτό και καλεί τη Βοσνία να απομακρυνθεί από το τέλμα και να κινηθεί και χτες στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών συζητήσαμε τη σημασία της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Αλβανία όπου ο Μύρος Λαβλάιτσεκ ως ε, δικός μου απεσταλμένος έχει αναλάβει να διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και την αντιπολίτευση. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, αν σκεφτούμε ευρύτερα το Σαχέλ και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε το Μαλί, τη Μαυριτανία, τον Νίγηρα και ευρύτερα το Μαγκρέμπ, ώστε να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα αναπτυχθεί μια προσέγγιση που θα διαφορεποιεί κάθε χώρα, αλλά θα, γενικά θα καλύπτεται από μια στρατηγική προσέγγιση σε ολόκληρη αυτή την περιοχή, ώστε να αντιμετωπίσουν ε, θέματα ασφάλειας, οικονομικά ζητήματα, ανησυχίες, ε, προβληματισμό όσον αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ναρκωτικών, θέματα που καθημερινά απασχολούν όλη αυτή την περιοχή και αν ε, κινηθούμε πιο κάτω στην Αφρική, στο κέρας Αφρικής, να μην εστιάσουμε μόνο στην πειρατεία που είναι βέβαια πολύ σημαντική, αλλά να δούμε και πώς θα στηρίξουμε οικονομικά τη Σομαλία, πώς θα δημιουργηθεί ηγεσία στην Αφρική και επισκέφθηκα την περιοχή δύο φορές, ώστε να έχουμε μια γενική εικόνα για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη να στηρίξει την περιοχή αυτή. Συχνά λέω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει μακροπρόθεσμα. Έργο μας είναι να οικοδομήσουμε τη βαθιά δημοκρατία, να στηρίξουμε τις χώρες που περνούν μεταβατική περίοδο και αλλαγές, να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά την κοινωνία των πολιτών, την πολιτική, την οικονομία τους, ώστε μακροπρόθεσμα να χαίρουν ε, δημοκρατικών θεσμών και οικονομικών προοπτικών και χρειάζεται μια υπηρεσία που να μπορεί αυτά να τα επιτύχει. Η, η ανάπτυξη χέρι με χέρι με την ασφάλεια, οικοδόμηση εμπιστοσύνη και θεσμών βαθιά δημοκρατία την οποία οικοδομούμε ε, λιθαράκι, λιθαράκι. Δεν είναι και πολύ ε, ένδοξα όλα αυτά, αλλά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να ενεργήσουμε πολύ αποτελεσματικά. Αν θέλετε, είναι σαν ένα μεγάλο τάγκερ, μια μεγάλη δεξαμενή που είναι η υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπηρεσίε τη, αλλά χρειάζεται ένα ταχύπλο που να μπορεί εύκολα να ελιχθεί σε δύσκολε περιστάσει, ώστε να στηρίξει ε, επιτόπου της χώρας και αυτό έχει τεράστιε επιπτώσει για το πώ ε, θα λειτουργήσει η εξωτερική υπηρεσία στο μέλλον λαμβάνοντα υπόψη ότι ακόμα βρισκόμαστε στη φάση τη οικοδόμηση, στην αρχή Τη δουλειά μα. Πρέπει επίση να σκεφτούμε από πολιτική άποψη και να βελτιωθούμε όταν ε, δρούμε σε πραγματικό χρόνο. Επίση θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ό,τι και αν κάνουμε, το κάνουμε σε συνεργασία με του εταίρους μα και γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε πολύ χρόνο και ενέργεια στι σχέσει κλειδιά που είναι τόσο σημαντικέ. με τα Ηνωμένα Έθνη και το Γενικό Γραμματέα με τον οποίο έχω συναντηθεί πολλέ φορέ και με τον οποίο συνομιλώ τακτικά. Επίσης ε, με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής, ε, το Χίλαρη Κλίντον και το επιτελείο της με την οποία συνομιλώ κάθε ώρα με τον Γενικό Γραμματέα Άμαν Μούσα της, του Αραβικού Συνδέσμου, με την Αφρικανική Ένωση, τον Σον Πίνγκ, με τον οποίο συζήτησα σήμερα, τον Γενικό Γραμματέα Ράσμουσεν του ΝΑΤΟ, με τον οποίο συνομιλούσα χτες, με τη Ρωσία, με την οποία έχουμε ένα μακρύ και βαθύ διάλογο με την Κίνα για την δουλειά που κάνουμε όχι μόνο στηρίζοντας μαζί με την Κίνα και άλλες χώρες για να δούμε πώς προσφέρουν πόρους ώστε να στηρίξουν την μετάβαση στην Τινησία και στην Αίγυπτα μαζί με πολλές άλλες χώρες που ήρθαν στην ε, Βρυξέλλες υπό τη δική μας προεδρία και με την Τουρκία που ίσως σε ορισμένε περιπτώσεις είναι ο πιο στρατηγικός εταίρος που έχουμε και με τον οποίο ε, διαρκώς ε, συνομιλούμε τακτικά με τον, Υπουργό Εξωτερικών Ταβούτογλου αλλά και Έχουμε ε, σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη στήριξη, με τον επιχειρηματικό κόσμο, μιλάμε με τις εταιρείες ε, παραγωγής ενέργειας που φυσικά ανησυχούν για το τι συμβαίνει με την πυρηνική ενέργεια με την ε, Ιαπωνία, αλλά και τι συμβαίνει στη Λιβύη και στο πετρέλαιο και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει δηλαδή διαρκώ να είμαστε σε επαφή με όλου σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον και ατζέντα για το μέλλον για να έρθω τώρα στην γειτονιά μας και να ξεκινήσω μετά της Λιβύης. Φυσικά τεράστια αλλαγή συνέβη όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας πέρασε το ψήφισμα 1973. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν σαφές ότι για να γίνει οτιδήποτε έπρεπε να υπάρχουν τρεις στόχοι. Νομική βάση, του Συμβουλίου Ασφαλείας στήριξη από την περιφέρεια και την Αραβικό Σύνδεσμο και τις ανάγκες του κόσμου. Αυτοί οι, τρεις, όροι, αν ε, πληρούνταν, θα έπρεπε να προβούμε σε δράση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο που εμείς πρέπει να παίξουμε και που συζητούσαμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εχθές και που υπήρχε ομοφωνία απόψεων, είναι σαφές όσον αφορά την ε, ουσιαστική φύση της ανθρωπιστικής μας στήριξης. Η δουλειά που ήδη έχουμε κάνει από τους 7.000 Ευρωπαίους που έφυγαν από τη Λιβύη, 4.400 έφυγαν με στρατιωτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να τους φέρουμε πίσω. Από τον κόσμο που περιμένει στα σύνορα, 20.000 άνθρωποι, κυρίως Αιγύπτιοι, ε, πολίτες του Μπαγκλαντές και άλλοι, έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους μέσω της δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κόσμο ακόμα στα σύνορα που στηρίζουν όσους φεύγουν από την Λιβύη και έχουμε στην Τρίπολη και στη Βενγάζη κόσμο που συζητά με το λαό για το τι συμβαίνει, έρχονται σε, ε, κάνουν επαφές ιδιαίτερα στη Βενγάζη για να κατανοήσουν ποια ακριβώς είναι η κατάσταση και για να εξετάσουν τι γίνεται όσον αφορά τα τρόφιμα, το νερό, τη φάρμακα. Ε, μιλάμε με τους ε, γιατρούς χωρίς σύνορα, με τον Ερυθρό Σταυρό, να δούμε τι υπάρχει και τι πρέπει να προετοιμάσουμε για την κατάσταση μετά την σύγκρουση και επανέρχομαι στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγώ πιστεύω βαθιά πως είναι να ε, βοηθήσει τις χώρες να προετοιμάσουν το μέλλον τους αλλά με ηγεσία των ίδιων των χωρών και για την Αίγυπτο και την Τινησία επισκέφθηκα την Αίγυπτο δύο φορές από την αποχώρηση του Μουμπάρακ. Ήμασταν οι πρώτοι μάλιστα που καλωσορίσαμε αυτή την αποχώρηση. Και άκουσα διάφορα μηνύματα και ξέρω ότι ο πρόεδρος Μπούζε και όσοι πήγαν στην Αίγυπτο το άκουσαν επίσης. Αυτή είναι η χώρα μας, είπε, είπε ο λαός της Αιγύπτου. Αυτή είναι η δική μας επανάσταση. Με τους νέους που συνάντησα στην ε, πλατεία Ταχρέκ, τους νέους ηγέτες του μέλλοντος είπαν ότι θέλουμε εμείς να εκλέξουμε τους ηγέτες μας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η φιλοδοξία τους και επίσης λένε ότι το σύστημα θα πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία αυτής της αλλαγής και χρειαζόμαστε βοήθεια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Αιγύπτια υπουργό Προγραμματισμού, μια γυναίκα εξαιρετικά δραστήρια, δουλεύει σε ένα πρόγραμμα για να ε, χτιστούν ε, καταλήματα για πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Θέλει να αναπτύξει αυτό το πρόγραμμα, να δώσει επίσης ε, κατάρτιση επαγγελματική για τους ε, νέους, να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βοηθήσει τον κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο και να ε, γίνει κάτι πια πραγματικότητα. Εγώ θέλω να τη βοηθήσουμε να γίνει αυτό. Θέλω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η BERD να δώσουν το μάξιμουμ των πόρων που γίνεται να συμμετέχουμε μαζί με όλες τις χώρες που μας ρώτησαν πώς να βοηθήσουν, να συντονίσουμε την προσέγγιση μας και να στηρίξουμε τον λαό της Αιγύπτου σε αυτή την προσπάθεια. Επίση γνωρίζουμε ότι στην Τινησία χρειάζεται στήριξη του Ζαν Πίνγκ της Αφρικανικής Ένωσης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Τινησία. Του μίλησα και μου είπε ότι ο λαός είναι πολύ αισιόδοξο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ήδη στην Τινησία έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα, αλλά πρέπει ακόμη περισσότερο να βοηθήσουμε ώστε να γνωρίζουν ότι δεν τους δίνουμε μόνο κάποια χρήματα όπως αυτά που τους έδωσα όταν πήγα εκεί, αλλά πρέπει να δούμε πιο μακροπρόθεσμα ποια θα είναι η στήριξή μας. Πρέπει αυτό να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Ε, θα πρέπει να επιθυμούμε και εμείς να πετύχουν αυτές οι μεταβάσεις και να δώσουμε τους απαραίτητους πόρους ώστε να ε, πετύχουν όντω. Και γι' αυτό και με την Κομισιόν κάναμε μια κοινή, ένα κοινό ανακοινοθέν μαζί με τον Πρόεδρο Μπαρόζο για να αναπτύξουμε αυτό που νομίζω ε, χρειάζεται και αυτό να το υποβάλουμε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κατ' ουσίαν είπαμε ότι υπάρχουν τρία πράγματα. Χρήματα, χρήματα, πόροι ε, η δυνατότητα να μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη μέσω των δικών μας προγραμμάτων και μέσω της ε, ανακατασκευής των προγραμμάτων μας ώστε να έχουμε ευέλικτους πόρους που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και επιπλέον να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και άλλους πόρους, είτε πρόκειται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μίλησα για την ΕΤΕ και την ΠΕΡΔ, υπάρχει Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι, αλλά και κράτη-μέλη. Δεύτερον, ε, πρόσβαση στην αγορά, να αρθούν τα εμπόρια, τα εμπορική φραγμή, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση μαζί μας και να αναπτυχθεί η οικονομία τους και τρίτον κινητικότητα. Ιδιαίτερα όταν σκεφτόμαστε τους νέους πληθυσμούς, το δυναμικό των φοιτητών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη σύνδεση μαζί μας και να καταστήσουμε ευκολότερη την κίνηση του, τη μετακίνηση του. Αυτό όμω θα πρέπει να το εφαρμόσουμε κιόλα. Να γράφουμε ένα έγγραφο εντάξει, αλλά πρέπει και να το θέσουμε σε εφαρμογή. Γι' αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει διεθνή συντονισμό που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό με χώρε σε ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν από την Τουρκία στην Αυστραλία, την Κίνα, τη Ρωσία ώστε όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την ε, περιοχή. Οπότε κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα φτιάξουμε τον κατάλληλο μηχανισμό που θα μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά, χρησιμοποιήσουμε τους πόρους σωστά και αποτελεσματικά, ότι θα Έχουμε επαφέ με του λαού ώστε να είναι ναι, η δική του επανάσταση και η χώρα του και η δική μα υποστήριξη θα κάνει ακριβώ αυτό θα του στηρίξει. Και επίσης θα καταστήσουμε σαφές ότι η δικιά μας δουλειά είναι να φτιαχτεί αυτή η βαθιά δημοκρατία και η βαθιά οικονομική ε, ανάπτυξη. Ε, να αισθανθούν ότι έχουν μακροπρόθεσμα ασφάλεια και ε, συνεργασία μαζί μας. Και έτσι λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ. Grazie, Ευχαριστούμε πολύ την ε, κυρία Άστον. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ε, παρέμβασή σας και διάβασα κάποια άρθρα του, κάποια κομμάτια αποσπάσματα του άρθρου στη New York Times σχετικά με την αγορά, τα χρήματα και την κινητικότητα στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με το πρώτο που είπατε, δηλαδή την χρηματοδοτική παρέμβασή μας στα κράτη για τα οποία μιλάμε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, πολύ σημαντικά ποσά που είναι απαραίτητα τόσο για εκτακτή ανάγκη όσο και για την οικοδόμηση υποδομής, για την επαγγελματική κατάρτιση και το καθεξής. Είναι λοιπόν δύσκολο να βρει κανείς αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της κρίσης, τόσο σημαντικά κονδύλια. Όμως, ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο να κατορθώσουμε να επιτύχουμε τη σωστή χρήση αυτών των κονδυλίων, να βοηθήσουμε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή ε, μπορούμε να βρούμε αξιόπιστους ε, εταίρους, αποτελεσματικούς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς, δηλαδή να δημιουργήσουμε την υποδομή της δημοκρατίας. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπάτη, εκπρόσωπε εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τόσο γρήγορα έρχεστε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών. Δεν θα ήταν ε, δίκαιο να σας ε, υποδεχθούμε σήμερα με νέα κριτική δοκιμάζονται οι δομέ τη συνδέξη Λισαβόνα από την κρίση που γνωρίζουμε αυτό το καιρό στην νότια όχθη τη Μεσογείου και στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας και των αρμοδιοτήτων σας ε, εργάζεστε καλά. Ε, συνεργαζόμαστε ε, καλά με τις υπηρεσίες σας. Εσείς έχετε υποβάλει μια φιλόδοξη ανακοίνωση και σωστά κάνετε μια διάκριση μεταξύ του βραχυπρόθεσμου, του μέσο και μακροπρόθεσμου ε, στόχου στην πολιτική γειτονία. Επίση, πολύ γρήγορα εφαρμόσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ψήφισμα 1970 πρώτα του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ. Καταφέρατε να Επεκτείνεται αυτή την εντολή και όπως ζητούσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκαλέσατε και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας γιατί ε, για αλλαγή δεν κινητοποίησαν όλη αυτή την κατάσταση οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η ε, Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με το Λίβανο που παρουσίασαν το σχέδιο ψηφίσματος 1973 στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μερικά σχόλια όμως κυρία Ήπατη, ε, εκπρόσωποι που ε, γεννούν και μερικά ερωτηματικά. Δεν φταίτε εσείς, αλλά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ακολούθησαν ε, την ίδια στάση στη ψηφοφορία. Το ίδιο ισχύει για το ΝΑΤΟ. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κυρία Άστον, για να βελτιώσουμε το συντονισμό μας σε αυτούς τους τομείς. Δεύτερον, Διάβασα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών εχθές, όπου εκφράζεται ε, την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εφαρμόσει το ψήφισμα 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γνωρίζουμε ότι βραχυπρόθεσμα δεν έχουμε δυνατότητα μόνοι μας να το κάνουμε αυτό ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να το πράξουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε λοιπόν κυρία Άστον τη λήψη των αποφάσεών μας, να γίνεται με ταχύ ρυθμό και επίση, μόλι επιστρέφουμε από την Αίγυπτο, ορισμένοι συνάδελφοι, ε, ήμασταν παρόντες στο δημοψήφισμα που τροποποίησε το Σύνταγμα. Διάβασα τη δική σα δήλωση για αυτό το δημοψήφισμα, αλλά θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Πώ αξιολογείτε πολιτικά εσεί το γεγονό ότι το 77% των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα ακολούθησαν τι συστάσεις τη μουσουλμανικής αδελφότητα και του παλιού. Ε, εκπροσώπους του κόμματος του κυρίου Μουμπάρακ σε αντίθεση με τα όσα συνιστούσαν οι κύριοι Μούσα και Μπάραντεϊ. Εσείς ε, πώς το αξιολογείτε αυτό. Το κοινοβούλιο ήταν πολύ επικριτικό κάθε φορά, ιδιαίτερα τελευταία, σε σχέση με κάποιες θέσεις που ακούγονταν και εκδηλώθηκαν από κάποια χώρα μέλος και προκειμένου τη Γαλλία. Θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να εκφράσω την αναγνώρισή σας την αναγνώριση γνώμη για ε, τη στάση της Γαλλίας απέναντι στη Λιβύη ε, για το στένος και την αποτελεσματικότητα υποστηρίζουν τους ε, αντιφρονούντες συγκάλεσαν τη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού και μία ώρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής άρχισαν να εφαρμόζουν το ψήφισμα. Μετά από όλες αυτές τις επικρίσεις που είχαμε εκφράσει τώρα θέλουμε να συγχαρούμε τη χώρα αυτή γιατί πραγματικά είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Mm, mm, συνάδελφοι, ε, θέλω να σας υπενθυμίσω και λυπάμαι που πρέπει να το κάνω αυτό, ότι στις 5 ε, πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ ε, να σέβεστε το χρόνο που σας προσφέρετε. Για τους συντονιστές είναι τρία λεπτά και δεν μπορούμε πια να δεχτούμε κανέναν άλλο να τον προσθέσουμε στην, στον κατάλογο των ερωτώντων γιατί σας είπα θα πρέπει να ε, τελειώσουμε στις πέντε. βηγαίνει επόμενος. Πρόεδρε, ε, θα προσπαθήσω να μιλήσω ένα λεπτό λιγότερο για να έρθουμε στα ίσα με το χρόνο που χρησιμοποιήσει ο κύριος Σαλαφράγκα. Κύριε Άστον, ε, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι ε, την ε, περασμένη εβδομάδα και το τελευταίο χρονικό διάστημα γενικότερα είχατε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσετε κι εσείς να κατανοήσετε τις δικές μας απόψεις και να καταρτήσετε τη στρατηγική σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, για ένα πολύ επίκυρο θέμα, προφανώς την κατάσταση στη Λιβύη. Τις τελευταίες εβδομάδες μιλήσατε για μια νέα ε, συνεργασία για τη δημοκρατία ε, και την ευημερία. Όμως δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, προτάσεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό αυτή τη στιγμή, πώς μπορούν να ιτηθούν οι δυνάμεις του Καντάφη. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να υιοθετήσει το ψήφισμα 1973. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς θα συμβεί. Και κατά τα άλλα, υπάρχει άραγε κάποια συζήτηση για να αποφευθούν τα λάθη του παρελθόντος ε, ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα, ποια είναι η στρατηγική εξόδου μετά από αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση και μετά την απομάκρυνση του Καντάφη που ευχόμετα. Την Κυριακή ο Αρμαμούσα, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, ανέφερε τρεις αρχές ε, και είπε ε, να μην υπάρξει εισβολή χερσαίων δυνάμεων, να υπάρχει προστασία του άμαχο πληθυσμού αυτό νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για την κατάρτιση της ε, στρατηγικής μας. Και ερωτώ τελικά, θα ζητήσετε την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση ή τουλάχιστον θα το συζητήσετε με τις Αιγυπτιακές Αρχές να δοθεί τέτοιου της βοήθεια. Γιατί από τότε που υπάρχει κατάσταση στη Λιβύη υπάρχει αποσταθεροποίηση και στην Αίγυπτο. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες της Αιγύπτου οι οποίοι ε, δεν θα μπορούν να αποστείλουν εμβάσματα και αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στην Αίγυπτο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει κάποια δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Αίγυπτο όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ ωραία. Κύριε Βιγγένιν, ε, στην άλλη κύριε Βιγγένιν, παράδειγμα προς αποφυγή, ε, Νέτς. Ευχαριστώ. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι, είπατε στην αρχή ότι από τον Οκτώβριο δεν έχετε έρθει φαίνεται ε, πολύ λιγότερο το διάστημα. Γι' αυτό σημαίνει ότι ήσασταν πάρα πολύ καλά εκπροσωπούμενοι εδώ, πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να σας βλέπουμε όσο γίνεται συχνότερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη γενική επισκόπηση που μας κάνατε, αλλά μια επισκόπηση που είναι πραγματικά ε, πολύ ζωφερή. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε συμβαίνει απανταχού της γης οποιοδήποτε θα είχε προβλήματα να τα ε, χειριστεί και να αντιμετωπίσει. Έρχομαι τώρα σε μερικά συγκεκριμένα ε, θέματα, κύριε εκπρόσωπε. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλήσατε για τη Λιβύη. Τονίσατε κυρίως την ανάγκη να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη εν γέννη. Αλλά όπως τόνισαν και προλαλήσαντες, αποσιωπήσατε τους πολιτικούς στόχους και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν αυτοί να επιτευχθούν. Βεβαίως, το Συμβουλίο Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ έχει ένα ψήφισμα το οποίο παραμένει και αυτό ασαφές και συγκεκριμένο για τον απότερο πολιτικό στόχο. Επίσης είπατε για την Τουρκία και σας παραθέτω ότι είναι από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους γενικότερα στην ευρωπαϊκή της Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, αλλά υπό το φως αυτό είναι περίεργο που η Τουρκία ε, ήταν απούσα από τη συνεδρίαση των Παρισίων. Και βεβαίως δεν σας ε, ζητήσω να το σχολιάσετε αυτό για τη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά ίσως να μας πείτε ποια είναι η προσωπική σας αίσθηση. Εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι κάνετε για να συμμετέχει πλήρως η Τουρκία στα όσα συνέβησαν και στα όσα συμβαίνουν και πρόκειται να συμβούν. Και να πω δύο λόγια για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, και εκεί έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο λέγουν ότι ε, το επόμενο διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ίσως θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ. Grazie. Collega Branner, prego. Ja, herzlichen Dank. Ähm, herzlich willkommen bei uns im σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Καταρχήν όσον αφορά τη Λιβύη. Ε, πρέπει να εκφράσω ε, τη λύπη μου ε, για το ότι είστε αναγκασμένοι να διαπραγματευτείτε με την γερμανική κυβέρνηση. Αλλά να ξέρετε ότι δεν συμφωνούμε όλοι με τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει το ότι η Γερμανία ακολουθεί το δικό της τον δρόμο. Βεβαίως γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει εσάς. Η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες χώρες ακολουθούν τον δρόμο τους και εσείς έχετε μία δύσκολη εποχή μπροστά σας. Η, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εφαρμόσει εμπάργο ε, και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτά κατά μέρο. Α πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι σωστά τοποθετηθήκατε στι χώρε εκείνε όπου ήδη έλαβε χώρα η Επανάσταση. Όμω δεν άκουσα να κάνετε σχόλια για τι χώρε εκείνε όπου αναπτύσσεται βία, όπου βράζει το καζάνι, με τι οποίε όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει ε, φυσιολογικέ σχέσει. Α πούμε, με τη Συρία. μήπω να να πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση μας απέναντι στη Συρία. Η Εμένη, 15 εκατομμύρια από το μέσο σταθερότητας χορηγούνται αυτή τη στιγμή στην Ιέννη ε, για μεταρρυθμίσεις. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε τη δουλειά που κάνουμε και να την αναξιολογήσουμε. Μαρόκο, Δυτική Σαχάρα, Συμφωνία Ελίας, ε, μπορούν να αναθεωρηθούν όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να μας δείξετε περισσότερο ότι δεν τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, αλλά αντιδρούμε εκ των προτέρων και ε, εξετάζουμε όλες τις ε, δυνατότητες. Και ένα άλλο θέμα. Αναφερθήκατε στην ε, Τράπεζα Νοικοδόμηση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμηση. Νομίζω πρέπει να προσέξουμε να δούμε ποια ήταν η εντολή μέχρι τώρα αυτή τη χώρα. Οι περισσότερε ε, χώρε συνέβαλαν στην ιδιωτικοποίηση και προέβαλαν πολιτικέ οι οποίε δεν νομίζω ότι έχουν καμία σχέση με την κοινωνική ειρήνη και την ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί για το μοντέλο που εξάγεται σε αυτέ τι χώρε και κατά πόσον οι χώρε επιτόπου ε, εποφελούνται. Και τέλος, ε, κώδικα ε, συμπεριφοράς σε σχέση με τα όπλα. Υπάρχει αυτός, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να χορηγούνται όπλα σε καθεστώτα όπως αυτό του Καντάφη. Ποια είναι τα προγράμματά σας για να είναι πιο αυστηρό το πρόγραμμα αυτό, να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα και με την πρωτοβουλία Transparency International που λέει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνειες χώρες που έχουμε σχέσεις για εισαγωγές πετρελαίου εσείς πώς ακριβώς αξιολογείτε αυτή την ε, τοποθέτηση. Τάνοκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, βεβαίω στην πολιτική μια εβδομάδα είναι πολύ μεγάλο διάστημα αυτό τον καιρό και δεν ήταν πάρα πολύ ένδοξη η για την ΚΕΠΑ και την ενότητά τη με τη γερμανική αποχή στο Συμβουλίο Ασφαλεία και την Τουρκία να χρονοτριβεί. Ε, και τώρα ε, μπορεί το ΝΑΤΟ να αναλάβει την επιβολή της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Κάνετε υπερορίες κυρία Άστον, το γνωρίζω και θα πρέπει να σας συγχαρούμε. Τώρα που μιλούμε για οικονομική σταθεροποίηση της Νότιας Μεσογείου σε ένα κλίμα μεγαλύτερης δημοκρατίας και των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, πιστεύω ότι η δική μου ομάδα σίγουρα θα υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο θα ήθελα να πω εδώ για τη Λιβύη, πέρα από το γεγονός ότι το 1973 δεν το επιτρέπει ε, ή δεν το αναφέρει. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει το καθεστώς, γιατί όσο επικρατεί ο Καντάφη δεν πρόκειται να υπάρξει δημοκρατία στη χώρα, γιατί την νησία... χάρηκα που έμαθα ε, ότι η ε, Φορευτική Επιτροπή ε, απαγόρευσε τη συμμετοχή δύο Ισλαμικών ε, κομμάτων ε, γιατί έχουν πολύ ανετικές τάσεις απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις γυναίκες. Στην Αίγυπτο παρά την επανάσταση που έγινε οι χριστιανοί, οι κόπτες και άλλες μειονότητες υφίστανται διακρίσεις και διώξεις βάρος τους με προσχήματα τη βλασφημία. Επίση, στο Μπαχρέιν, τη Συρία και στην Ιεμένη έχουμε νέε εξελίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα πρέπει να έχει διπλέ ε, ε, Αρχέ, δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα πρέπει παντού να πρεσβεύει τα ίδια. Επίση δεν θα πρέπει να ξεχνούμε του ανατολικού γείτονε. Τώρα έχουμε στραφεί προ τον νότο και έχετε υποσχεθεί εδώ και καιρό ότι θα πάτε στο Κίεβο να επισκεφτείτε το στρατηγικό μας εταίρο την Ουκρανία που κινδυνεύει ε, να ε, στραφεί γεωπολιτικά αλλού, όχι προς τη δική μας κατεύθυνση. Και σε ό,τι φορά τη ε, Ρωσία και τα σχόλια του Πούτιν για τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που τη χαρακτήρισε σταυροφορία. Διαφώνησε με τον Μετβέντεφ, ο οποίος τον κατατρόπωσε. Τι έγινε αυτό το δίδυμο εκεί, έχει αρχίσει να σπάει στο Κρεμλίνο. Ευχαριστώ. Κολέγα Μέιερ, ο συνάδελφος ε, Μάιερ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, γνωρίζετε ότι η πλειοψηφία τη ομάδα μου είναι απολύτω αντίθετη με την ξένη επέμβαση για να λυθεί ε, η κατάσταση και η σύγκρουση στη Λιβύη. Εμεί συμμεριζόμαστε τα μελήματα και τι ανησυχίε που οδήγησαν τη ε, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Γερμανία στην αποχή σε αυτό το ψήφισμα. Διότι πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν ε, στρατιωτικά ε, να επιβληθούν. Έχουμε πάνω από 32 τέτοιες καταστάσεις σε χώρες στον κόσμο. 32. Κανείς δεν θα είχε αυτή την ε, τρελή ιδέα να κάνει στρατιωτική επέμβαση και κανείς δεν ξέρει πού το πάμε. Ορισμένοι λένε να πέσει ο Καντάφη και αμέσως τους διαψεύδουν. Άλλοι λέγουν ότι ηγείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την προσπάθεια και διαψεύδεται αμέσω μετά. Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ και πάλι δεν βρίσκει την απαραίτητη πλειοψηφία για να αποφασίσει εάν ε, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναλάβει τη διοίκηση. Και τέλος, αποκλείεται ε, στρατιωτική κατοχή χερσαία και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου γίνονται επιλεκτικοί βομβαρδισμοί με πυράβλου κρού που δεν κάνουν διάκριση οι πύραυλοι που θα πάνε και τι θα καταστρέψουν, αν θα είναι άρμα μάχη ή αν δίπλα έχει τον άμαχο. Και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι και ειλικρινά ο, ο Μπάνκι Μουν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα πρέπει τώρα να ε, μεταβεί εκεί να επιβάλλει κατάπαυση του πυρός και να αναγκάσει ε, τα αντιμαχόμενα μέρη σε διαπραγματεύσει. Πήγα και εγώ με τον κύριο Σαλανφράκα και άλλου συναδέρφου στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι ρόλο έχει παίξει στην ε, Αφρική το 19ο και 20ο αιώνα η Ευρώπη. Και η αίσθηση που έχουν οι Αφρικανοί για οποιαδήποτε ξένη επέμβαση ευρωπαϊκή, προκειμένου στην Αφρικανική Ήπειρο. Μέχρι και ο Αραβικός Σύνδεσμος που έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ήδη ζητάει να σταματήσει αυτή η κατάσταση που ε, προχωράει πέρα από την καταστροφή των αντιαεροπορικών ε, δυνατοτήτων και της ε, δυνατότητας διαβιβάσεων πληροφοριών. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ την εντολή. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να τερματιστεί τώρα αυτή η κατάσταση. Βεβαίως, η υποχρέωση να παρέμβει κανείς για να διαπιστώσει την ε, κατάπαυση του πυρός. Αλλά έχουμε σε ύψιστο αξίωμα τον κύριο Μπάνκι Μουν και του ζήτησε και ο Λούλα, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, να μεταβεί ο κύριος Μπάνκι Μουν και να τους υποχρεώσει να διαπραγματεύονται με κατάπαυση του πυρός η οποία να αποδεικνύεται. Και να σταματήσει αυτό ε, της διγλωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκατάφη που δεν αξίζει τον παραμικρό σεβασμό από τη Δημοκρατική ήταν στενό φίλο Μπερλουσκόνη Σαρκοζή τη κυρία Μέρκελ και όλων των Ευρωπαίων ηγετών. Και δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη από την εγκάρδια φιλία να περάσει κανείς στην έχθρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κλείσει λοιπόν τον ε, πρώτο ε, γύρο των ερωτήσεων που υποβάλλουν στον Ιδέα, συνάδελφος κύριος Μπέλνε. Ο Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Άστον, είχα την ικανοποίηση και το προνόμιο τις τελευταίες μέρες να μεταβώ στην Αίγυπτο με την προσωπία του Κοινοβουλίου, όπου και εσείς οι ίδια πήγατε επανειλημμένα. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά ε, την ευρωπαϊκή βοήθεια ε, για τη στέγαση. Πάνω από 100.000 Αιγύπτιοι ζουν σε νεκροταφεία, σε καταστάσεις ανίποτες. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αναλφαβητισμού ε, μεταξύ των ενελίκων 24% παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει και το θεωρώ τεράστια σημασία. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ακούσαμε και διπλωμάτες και εσείς φαντάζομαι που μίλησαν για προβλήματα τρομερά ε, ε, οικονομικά και επισητιστική κρίση. Συμφωνείτε και εσείς η διαδικασία του ε, εκδημοκρατισμού κινδυνεύει να απειληθεί ε, από ε, αυτή την κατάσταση. Επίσης, είναι μεταβατική η περίοδος και ο στρατός έχει τεράστιο ρόλο. Μας διαβεβαιώνουν ότι είναι και αυτό μεταβατικό, αλλά το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές, εάν παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς, θαυμάσια. Αλλά αν ταυτόχρονα διατηρήσουν και μια οικονομική αυτοκρατορία ή στρατιωτική, πώς θα επέλθει το κράτος δικαίου ε, και πώς θα ανανεωθεί η κοινωνία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Grazie. La, la parola mh, mm, alla baronessa Ashton per le risposte. Colleghi, θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Άστον για να απαντήσει και συνάδελφοι θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στις παρεμβάσεις σας σε 1,5 λεπτό γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τον λόγο σε όλους όσοι τον έχουν ζητήσει. 1,5 λοιπόν λεπτό, το πολύ μία-δύο ερωτήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν τον λόγο όλοι και νομίζω αυτό είναι θέμα και δικαιοσύνης και ισότητας απέναντι στους συναδέλφους. Ε, πόσο θέλετε να μιλήσετε, μισή ώρα? Ξέρω ότι το είπατε για στείο το μισή ώρα. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και αναφερθώ ε, σε όσο το δυνατόν ε, περισσότερες ερωτήσεις. Εσείς με ρωτήσατε πρώτος σχετικά με την οικονομική παρέμβαση, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για με ρωτήσατε σχετικά το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα κονδύλια και από πού θα τα πάρουμε. Το θέμα είναι συνδυασμού πόρων που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να δούμε πώς μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα αναδιατάξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπατε κι εσείς ε, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα δαπανώνται σωστά και τομείς όπου υπάρχει υποχρηματοδότηση εκεί να σημειώσουμε κάποια βελτίωση. Εγώ νομίζω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα δις στην περιοχή αυτή. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος έχει 484 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ μεγάλο ποσό και η Τράπεζα Ανασυγκρότησης ε, και αυτοί ε, προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερα κονδύλια. Δεν θα αφαιρέσουν κονδύλια από την, τους ανατολικούς εταίρους μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζονται ακόμα βοήθεια. Και βέβαια και ο Μποπ Σέλιχ από την Παγκόσμια Τράπεζα και αυτό θα εμπλακεί. Άρα δηλαδή η δική μας πόρη και των υπόλοιπων οργανισμών σας ανέφερα. Κύριε Σαλαφράγκα, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πράγματι προσπαθούμε να αναδιαρθρώσουμε την πολιτική γειτονία, να είναι πιο αποτελεσματική, περισσότερο σε θέση να ανταποκρίνεται. Ο κύριος Φίλου. έχει κάνει πολλή δουλειά, ε, βεβαίω ε, υπολείπονται ακόμα πολλά, όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα και πολύ χρήσιμα. Ε, το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας, τα κράτη-μέλη και συντονισμός. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ακριβώς ο συντονισμός, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε 27 διαφορετικά κράτη-μέλη με εθνική κυριαρχία που είναι παθιασμένα ότι έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν μόνο τους ε, σε θέματα άμυνας και γι' αυτό και υπάρχει και ε, διαφορά απόψεων. Το θέμα όμως είναι ότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας κανείς δεν καταψήφισε το ψήφισμα. Και χθε επιτύχαμε ομοφωνία στο Συμβουλίο Υπουργών για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το βέλτιστο δυνατό τρόπο να βοηθήσει με ανθρωπιστική βοήθεια, με την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Νομίζω λοιπόν εδώ βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Ίσως ε, να μην είναι το καλύτερο, αλλά εκεί βρισκόμαστε. Και ο δικός μου ρόλος είναι να επιτυγχάνω, να προωθώ την ομοφωνία και να προβαίνω σε δράσεις. Όσον αφορά το δημοψήφισμα, ξέρω ότι και εσείς έχετε μελετήσει το θέμα και θέλω να πω το εξής. 42% είχαμε προσέλευση, μεγαλύτερη από ό,τι κατά το παρελθόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους Αιγύπτιους και στο αποτέλεσμα του μίλησε Μίλησα με τον κύριο Μπαραντάη ε, και με άλλου ε, και οι δύο γνωρίζουν ότι είναι υποψήφοι στις ε, προεδρικές εκλογές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για αυτούς να πιέζουν προ τα εμπρό. Αυτό σημαίνει εξάλλου δημοκρατία. Στην Αίγυπτο πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και του θεσμού. Και νομίζω μία από τι συζητήσει πολύ σημαντική για μένα στην Αίγυπτο ήταν πόσοι από αυτούς που συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία επιθυμούν να έχουν χρόνο για να είναι έτοιμη η πολιτική διαδικασία. Ε, υπάρχουν πολλοί εδώ με εμπειρία που ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να έχουν χρόνο τα πολιτικά κόμματα για να εξελιχθούν. Αυτό το επισήμανα. Ε, για μένα λοιπόν ε, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον. Ρωτήσατε επίσης ε, για, τις, ε, για τη δράση που πρέπει να αναλυφθεί απέναντι στον Καντάφη και το δρόμο που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, έβαλε τρεις όρους και όρισε κατά κάποιον τρόπο τις δράσεις. Η δράση λοιπόν που έχει αναλυφθεί ανελήφθη μετά από αυτά τα συμπεράσματα που εξήχθησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Για μας λοιπόν, εκείνο που παίζει ρόλο είναι να προσφέρουμε υποστήριξη στον άμαχο πληθυσμό. Και εδώ υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Σήμερα τα στρατεύματα του Καντάφη έχουν εστιάσει την προσοχή του σε μια πόλη 50 χιλιόμετρα μακριά από την Βεγγάζη, όπου είναι και η βασική ε, παροχή υδροδότησης ε, στην Βεγγάζη. Όπως είπα και προηγουμένως ε, στους αντέλφους, ε, στείλαμε ανθρώπους στη Βεγγάζη για να εξετάσουν την κατάσταση από πλευρά ε, εφοδιασμού τροφίμων και νερού. Ίσως χρειαστεί να υπάρξει κάποια απομάκρυνση πολιτών Πάντως μέχρι την πέμπτη αυτής της εβδομάδας θα είμαστε έτοιμοι και μετά θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Και αυτά πρέπει να τα συντονίσουμε με το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ συναντήθηκε σήμερα το πρωί, μόλις ε, τελείωσαν τη συνάντησή τους ε, και εξ όσων άκουσα, από αυτά που άκουσα, ε, θα συνεχίσουν το σχεδιασμό τους και θα μιλήσω κι εγώ αργότερα μαζί τους. Είναι δύσκολος ο διάλογος με τον Αμαμούσα. Πριν έρθω στη συνάντηση μίλησα μαζί του. Είναι σαφής, βεβαίως, αν δει κανείς το ψήφισμα των 1973 των ΗΠΑ είναι ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα. Την Πέμπτη θα υπάρχει συνάντηση ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο υπαριθμών 1 το 1 εκατομμύριο των ε, Αιγυπτίων ε, που δεν θα στείλουν εμβάσματα. Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι σημαντικό. Ε, εξετάζουμε το θέμα ευρύτερα. Τους τελευταίους μήνες έτσι κι αλλιώς από πλεόνασμα περνάμε σε έλλειμμα στην Αίγυπτο και πάρα πολλοί υποφέρουν γιατί ο τουρισμός ε, δέχθηκε ράπισμα από αυτά που έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στην Αίγυπτο. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αλλά και εκείνοι πρέπει να μας πούνε τι θέλουν, πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να συνεργαστούμε μαζί τους. Κυρία Νέιτς, η ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, συμφωνώ. Η πολιτική μου στόχη είναι πάρα πολύ απλή, νομίζω τους ανέφερα. Επιθυμώ οι κάτοικοι της Λιβύης να μπορούν να ορίσουν μόνο τους το μέλλον τους, δημοκρατία, ασφάλεια, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, από τους ε, εκπροσώπους τους ε, άκουσα ότι επιθυμούν να έχουν, έχουν δημοκρατία, να εκλέγουν τους εκπροσώπους. Αυτά που υπάρχουν εδώ στην Ευρώπη, μα είναι και οικουμενικές αυτές οι αξίες. Αυτά θέλουν. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Με την Τουρκία συνεργαζόμαστε συνεχώς. Ο κύριος Ομπάμα, ο πρόεδρος, ε, μιλάει με τους Τούρκους, τους μίλησε χθε το βράδυ. Εγώ μίλησα και μιλάω σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Πολύ σημαντικό αυτό για μας γιατί οι Τούρκοι είναι σημαντικοί εταίροι. Μιλήσαμε με ε, με τους, Τόρκους, ε, με τους Τούρκους και κάνουμε πολλή δουλειά στην Βοσνία και Σεγοβίνη. Συνεργαζόμαστε μαζί τους πάρα πολύ. Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πάρα πολλά, δύο-τρία θα πω. Πρώτον, πρέπει να μετακινηθούμε οπωσδήποτε. Το είπα και στους Ισραηλινούς ε, και στην Παλαιστινιακή Αρχή. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Μου είναι απόλυτα σαφές ότι στη γειτονιά αυτή είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια λύση. Ξέρουμε τα προβλήματα, ελπίζουμε να υπάρξει πρόοδος. Σύντομα θα έχουμε τη συνάντηση της ε, τετραμερούς. Ελπίζω η τετραμερής ε, να εκδώσει μια κατηγορηματική ανακοίνωση. Κυρία Μπραντνα, ο προγραμματισμός για το μέλλον. Μιλήσατε για τη Συρία. Μπορώ να φέρω Συρία, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Δυτική Σαχάρα. Ξέρω ότι η Επιτροπή Αρμόδια για την Αλία αναζητά και ψάχνει το θέμα, βρήκε μια ενδιάμεση λύση. Αυτό που κάνει ο βασιλιάς του Μαρόκου είναι πολύ σημαντικό και ένας τρόπος για να προχωρήσει η χώρα του. Ε, στο Μπαχρέιν, μόλις είπε τον Προκούπα από το Μπαχρέιν εχθές ε, το πρωί. Δικός μου ήταν ε, ο απεσταλμένος που πήγε στο Μπαχρέιν για να μιλήσει για την ψυχραιμία και για τον διάλογο που ξεκίνησε ο διάδοχος με κάποιες προϋποθέσεις. Η Συρία. βλέπουν και εκείνοι και είναι σημαντικό ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές και νομίζω αποκρίνονται Και έχετε δίκιο, πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτές τις χώρες, γιατί πιστεύω ότι ε, πρέπει τα προγράμματά μας ε, να αναγνωρίσουν τις αλλαγές. Αλλά ε, δεν δέχομαι αυτό που είπατε ότι υστερούμε, αλλά όχι. Τώρα είμαστε μπροστά. Μερικές φορές αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πράγματα που ίσως να ήμασταν πιο πίσω, αλλά τώρα είμαστε στην πρώτη γραμμή, πρωτοπόροι. Κύριε Τάνοκ, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Το ένα, της θρησκευτικής ανοχής ε, και της βίας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό ε, το έφτιαξα με τον ε, Τατάουι. Μιλήσαμε για την βία και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα και είναι σημαντικό οι άνθρωποι με όλες τις τα θρησκευτικά πιστεύω να προστατεύονται. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Εγώ το έχω κάνει ήδη ε, ξεκάθαρα στην Αίγυπτο και όπως και εσείς πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ως προς την Ουκρανία πράγματι έχουμε σχέση με την Ουκρανία. Θα τους επισκεφτώ σύντομα. Ε, τους έχω μιλήσει αρκετά και θα τους επισκεφτώ. Όμως και εκείνοι πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις ε, στη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών. Η μπάλα είναι στο δικό τους το τερέν. τώρα, ο κύριος Μπανκιμούν ανέκαθεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική διαδικασία. Ε, το ψήφισμα αναφέρει πολλά και εκείνος επιθυμεί να δει ε, την ε, πολιτική διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα για τους ανθρώπους. Δεν είναι αντίφαση αυτά που λέει, όπως σας είπα θα του μιλήσω και αργότερα και δεν νομίζω και δεν δέχομαι ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όμως το έχω πει και κατά παρελθόν. Πρέπει κανείς να αποφασίσει ανάμεσα στην συμμετοχή και στην απομόνωση. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με χώρες ε, που μπορούμε, από το πάντα είναι καλύτερο. Ε, υπάρχουν όμως και καθεστώτα που δεν το θέλουμε. Μερικές φορές απομονώνουμε χώρες γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά ξεκινάει κανείς από την αρχή ότι καλύτερη συνεργασία και φτάνει κανείς στην απομόνωση όταν πια δεν γίνεται. Κύριε Μπέλντερ, τα θέματα της ε, στέγασης, ε, οι άνθρωποι είναι στους δρόμους, όλα αυτά τα θέματα της στέγασης ε, και των τροφίμων είναι πολύ σημαντικά και εντάσσονται στο διάλογο που έχουμε τώρα με την Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος, πρώτο, πρώτη παρέμβαση συνάδελφος Μποντή και μετά κυρία Ντεκαϊδέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατικπρόσωπε. Οι αραβικές επαναστάσεις μας επιβάλλουν ε, φυσικά να αναθεωρήσουμε την πολιτική γυρνίαση ε, μας. Ελπίζουμε μέσω αυτού του εργαλείου να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και φαίνεται πως πολύ συχνά έχουμε χρηματοδοτήσει αυταρχικά ε, καθεστώτα Τώρα, για να μην επαναληφθούν αυτά τα σφάλματα, είμαστε σε πλήρη αναθεώρηση της πολιτικής γετνίασης. Ο κύριος Φούλε μας έστειλε τα σχετικά έγγραφα. Το ερώτημα που εγώ έχω να θέσω είναι, τι κάνουμε απέναντι σε χώρες που είναι μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική γετνίασης, αλλά των οποίων το αυταρχικό καθεστώς παραμένει στη θέση του. Τι κάνουμε με μια χώρα γείτονα με την οποία συνδεόμαστε που καταστέλει και πνίγει στο αίμα τους επαναστάτες, τους διαδηλωτές. Θα ήταν δηλαδή καλό να προχωρήσουν οι συμφωνίες με τις χώρες των οποίων έχει αλλάξει το καθεστώς για να προχωρήσει προς τον ε, εκδημοκρατισμό, αλλά τι κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις. Προβλέπουμε αναθεώρηση όλων των συμφωνιών σύνδεσης που είναι ενισχύ με τους νότιους γειτονές μας. Ευχαριστώ. Άλλο υπόδειγμα σύνθεσης και συνοπτικότητας. Κυρία Ντικέζερ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωποι, επιτρέψατε μου με τη σειρά μου να σα συγχαρώ για τι ε, δράσει σα και για τη δράση τη υπηρεσία σα στο πλαίσιο των ε, Αραβικών Επαναστάσεων καθώ και για την δέσμευσή σα, Ευχαριστώ επίση τι υπηρεσίε σα που μου έστειλαν μια επιστολή με συμπληρωματικέ πληροφορίε για την τελευταία συνεδρίαση τη Συμφωνία Σύνθεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ. Έχω δύο ερωτήσεις σήμερα. Γνωρίζετε σε ποιο βαθμό σας στηρίζουμε για να σας βοηθήσουμε να αποδείξετε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι πραγματικά μια προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Υπάρχουν δύο τομείς όπου έχω κάποιες μικρές, ε, μικρούς προβληματισμούς. Πρώτον, η κρίση στην Ιαπωνία. Κρίση στην Ιαπωνία όπου τουλάχιστον ε, από εξωτερική άποψη φάνηκε να μην υπάρχει συντονισμό ανάμεσα στα κρατη τόσο όσον αφορά τι έπρεπε να γίνει, όσον αφορά επίσης τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν, ε, τι πρέπει να κάνουμε με τους ε, πολίτες μας εκεί, τους Ευρωπαίους ε, πολίτες, το ιόδιο, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πυρηνικό ατύχημα, πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίστηκε, αν το κατάφερε να συντονιστεί, και τι δίδαγμα αποκομίζεται από αυτή την αντιμετώπιση της ιαπωνικής κρίσης. Δεύτερος προβληματισμός μου σχετίζεται με την, το Νότιο Σουδάν. Ε, θα προσπαθήσω να συνοψίσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, Νότιο Σουδάν, όπου φαίνεται ότι η μετάβαση προς την δημοκρατία δεν γίνεται τόσο ομαλά όσο ελπίζαμε και όπου μέσω αυτού του σχεδίου συντάγματος που θα πρέπει να συνταχθεί τώρα, ο πρόεδρος Αλβακύρ δεν ανοίγει τόσο όσο θα θέλαμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αντίθετα προσπαθεί να δρομολογήσει ε, την αλλαγή υπέρ του κόμματος του. Υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, είναι πολύ ε, πολύ προφανή τα πράγματα και πώς θα θέλατε εσείς να συνοδεύσουμε αυτή τη μετάβαση προς την ε, ε, αλλαγή προς τον εκδημοκρατισμό. Κύριε Σπρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Άστον για την ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου ε, σχετικά ε, με ε, την εταιρική σχέση και την πολιτική γειτονία ε, με την νότια όχθη της Μεσογείου. Στο Κοινοβούλιο έχουμε εγκρίνει πολλά ψηφίσματα και ζητάμε σαφή κριτήρια για να δίνουμε σε κάποιον ένα προηγμένο καθεστώς. Στο προσεχές μέλλον θα μας ενημερώσετε με τρόπο σαφή για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμστορ. Καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι με εκπλήσει το γεγονός ε, ότι οι πράσινοι πολύ χαλαρά παίρνουν αυτά τα θέματα της στρατιωτικής επέμβασης. Μετά από δεκαετίες ε, ε, ειρηνισμού έχουν αλλάξει τώρα τακτική. Και την Πέμπτη και, τα περασμένες, και τις περασμένες ημέρες θα μπορούσαν τα κράτη να είχαν συντονιστεί καλύτερα. Ε, η αναγνώριση των εξεγερμένων στη Βεγγάζη από τη Γαλλία ήρθε εξίσου χωρίς συντονισμό, όπως και η στάση στην ψηφοφορία. Ε, εχθές το Συμβούλιο ομόφωνα καλωσόρισε ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, επί τη βάση αυτή θα πρέπει να εργαστούμε και δήλωσε το Συμβούλιο ότι οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να υποστηριχθούν και να εφαρμοστούν με διαφοροποιημένο τρόπο. Σωστό είναι αυτό και έχει να παίξει το ρόλο του κάθε κράτος μέλος. Βαρώνει, ας τον έχω δύο-τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις στα αγγλικά. Πρώτη, ε, στείλατε ένα εκπρόσωπό σας στη Βενγάζη. Σε τι κατέληξε. Στη συνέχεια, ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον Μπαχρέιν είναι πραγματικά εντυπωσιακά, εκπληκτικά, για να μην πω ότι ενοχλούν, γιατί τηρούν ίσες αποστάσεις και από το καθεστώς και από τους διαδηλωτές και ε, τους καλούν σε συγκράτηση. Μα πώς μπορεί κανείς να κατηγορεί τους διαδηλωτές που διαδηλώνουν για τη δημοκρατία. Δεν ξέρω τι να πω. Η κυρία Λούνατσα για να απαντήσει για αυτά που είπατε περί ειρηνιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα Βαλκάνια, αλλά να πω κάτι ε, για τη διαδικασία με την κυρία Άστον, τον κύριο Βημό και άλλους από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην επικοινωνία με το Κοινοβούλιο για την κατάσταση και την κρίση στη Βόρεια Αφρική. Θέλω πραγματικά να εκφράσω την αναγνώρισή μου. Ήταν καλός ο τρόπος και βελτιώνεται η επικοινωνία. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα Βαλκάνια. Το πρώτο, σύντομο για τη Βοσνία Πότε σκοπεύετε να ορίσετε εκεί τον νέο επικεφαλή τη αντιπροσωπεία, γιατί από πέρσι τον Ιούνιο χειρεύει η θέση. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, απαραίτητο να έχουμε εκπρόσωπο εκεί. Και για το διάλογο Κωσόβου-Σερβία που είπατε και ίδια ότι είναι σημαντική διαδικασία, συμφωνώ και ελπίζω να πετύχει. Για πρώτη φορά μετά από τη δήλωση της, ε, την αρκή εξαρτησίας του Κωσοβού πριν από τρία χρόνια, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και διαπραγματεύονται εκπρόσωποι και των δύο για τη βελτίωση των πολιτών. Έχουμε πρόβλημα στο Κωσυφοπέδιο, όμως πήγα εκεί την περασμένη εβδομάδα και έχουν την αίσθηση ότι ο μόνος κερδισμένος από αυτή την υπόθεση τελικά θα είναι η Σερβία. Εσείς τι κάνετε. Δεν θα πρέπει να αρχίσει ο διάλογος για τη θεώρηση διαβατηρίων για να πιέσουν στο εσωτερικό ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσει η κυρία Μάστον και να αρχίσει αυτό το διάλογο και τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν έτσι ώστε να πιστέψουν και πάλι οι Κωσοβάροι ότι η Ένωση τους θέλει στους κόλπους της. E Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δηλαδή, Άστον, νομίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο σας επειδή έχετε και βασικές διαφωνίες μέσα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και ανάμεσα στα κράτη-μέλη, πράγμα που αναπόφευκτα θα ακολουθήσουν τις δικές τους ε, πορείες ανάλογα με την κυριαρχία τους και τις επιθυμίες τους. Φυσικά εσείς γνωρίζετε το βρετανικό σύστημα. Μήπως θα ήταν ε, λογικότερο να ορίσετε ε, καμιά δεκαριά υπουργούς, υπουργούς ε, να ασχολούνται με τα καθημερινά ζητήματα έτσι ώστε εσείς να εστιάζετε την προσοχή σας σε αυτά που είναι τα πιο πιο ουσιαστικά θέματα. Μέση Ανατολή, αυτό που γίνεται στην Γάζα και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται οι Ισραηλινοί είναι πραγματικά ντροπή. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν την ίδια άποψη. Τώρα, δεν πιστεύετε πως είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να ενθαρρύνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει παίκτη πλέον και όχι απλώς πληρωτής εκεί στις ε, διασκέψεις αυτές ώστε να λυθούν κάποιες από τις ε, δυσκολίες. Παντζέρη. Για τον χρόνο να μην σχολιάσω, μόνο ένα σχόλιο να κάνω. Δεν διαφεύγει κανένα η ανάγκη να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή δράση. Αντίθετα, έχουμε δράση των θελοντών βασικά. Ε, είναι βασική η διαφορά αυτή. Πρώτη ερώτηση. Πλήρης εφαρμογή του 1973. Όμως, αν ξεπεραστεί αυτό το ψήφισμα, τι θα κάνει η Ευρώπη. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή δράση μάλλον τι είδος ευρωπαϊκή δράση σκοπεύετε να θέσετε σε εφαρμογή για να ανακτήσουμε για να ε, μετριάσουμε αυτή την διαφορά όσον αφορά την ηγεσία αυτών των ε, ε, των επιχειρήσεων. Έπειτα, για τον ΟΗΕ δεν είναι πολύ πιστική η ιδέα ενός μοναχικού πρωταγωνιστικού ρόλου. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να ανακτήσει αυτή την πτυχή. Και έπειτα, στο Παρίσι δεν είδαμε την Αφρικανική Ένωση ε, κατά κάποιο τρόπο ήρθε, αλλά τελικά αποσυνδέθηκε από την παρέμβαση. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντική η σχέση με την Αφρικανική Ένωση, γιατί είναι επικίνδυνο να θεωρηθεί αρνητική και να, να θεωρηθεί αρνητικά αυτή η παρέμβαση και να, οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε μάλλον σε ένα σωρό προβλήματα. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να διατηρήσετε τις επαφές με αυτές τις δύο σημαντικές, τα δύο σημαντικά όργανα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χάουταλα που είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δύο πράγματα έχω να πω. Μου αναφέρθηκε ότι υπάρχουν κάποια πολύ δραματικά γεγονότα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορε χώρε. Ιδιαίτερα με ανησυχεί το τι συμβαίνει στη Συρία αυτή τη στιγμή. Φαίνεται πω 20.000 άνθρωποι έχουν ε, κατέβει σε διαμαρτυρία ε, κατά τη δολοφονία από τι ε, υπηρεσίε ασφαλεία δύο ανθρώπων και στην κηδεία οι κυβερνητικέ δυνάμει του καλωσόριζαν με δακρυγόνα. Πώς θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Φαίνεται να αντιμετωπίζουμε σε ορισμένε χώρες, τις ε, αραβικές χώρες, τόσο στην Αμέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Μήπως όντως πρέπει να αναθεωρήσουμε τις ε, πολιτικές μας απέναντι σε αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα. Κυρία Άστον, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πείσει τη Συρία ότι πρέπει να σταματήσει να καταπιέζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της. Δεύτερον, κυρία Άστον, θα με ενδιαφέρει πολύ να μας πείτε δύο λόγια να μας πείτε με δύο λόγια πώς αυτό το νέο Citizen, το κέντρο ε, κατάστασης είναι, ε, θα λειτουργήσει. Φαίνεται να είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής υπηρεσίας, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τι ακριβώς ρόλο θα παίζει σε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, δύο τελευταίες παρεμβάσεις στο δεύτερο γύρο είναι ο συνάδελφος Μαντλένερ και Κάμπελ. Ο κύριος Μαντλένερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Άστον, εσείς ε, βέβαια εξωτερική πολιτική. Ποια είναι, ποιο, ε, σε ποιον πρέπει να τηλεφωνήσει κάποιος για να μιλήσει για την εξωτερική πολιτική, όχι σε εσά σίγουρα. Στον κύριο Σαρκοζή, στον κύριο Κάμερον. Έχει εξαφανιστεί τελείως η ε, σημασία σας, φανήκατε τελείως περιττή. Οι, οι επισκέψεις σας μπορεί να είναι συχνές και πολλές, ε, αλλά τελείως ασήμαντες. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει. Γάλλοι, Γερμανοί, Άγγλοι, Ολλανδοί, εσείς δεν έχετε καμία σημασία. Σας έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις. Δεν είμαι μόνο εγώ εκείνο που θρυνεί, αλλά και οι φορολογούμενοι των καθαρών συνεισφορέων που πληρώνουν δισεκατομμύρια οι Ολλανδοί οι φορολογούμενοι ένα σωρό πεταμένα λεφτά για τη θέση σας που δεν έχει καμία σημασία και καμία αποτελεσματικότητα. Για την Αφρική είπαμε, για την Ιεμένη αναλαμβάνουν από ό,τι φαίνεται οι Ισλαμιστές, τρομοκράτες και μπορεί να το κάνουμε Αφγανιστάν στην Ιεμένη βάση από όπου θα ε, ε, ε, εκδράμουν και θα κάνουν τις επιδρομές τους οι τρομοκράτες. Και τι γίνεται με τη βαρβαρότητα στη Βόρεια Αφρική. Είναι φοβερό το φανατικό, το φασιστικό Ισλάμ που επελάβνει, πώς θα καταφέρουμε να τους κρατήσουμε εκτός της κυβέρνησης και πώς θα καταλάβει ο κόσμος ποιον μπορεί να εκλέγει, ότι μπορεί να εκλέγει τους ηγέτες τους. Ελπίζουμε να μην επικρατήσουν ε, οι φοβεροί, ε, φανατικοί, ε, φασιστές, Ισλαμιστές ηγέτες. Ο κύριος Κάμπελ στην τελευταία ολομέλεια η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης ε, έχει το ίμιση του ε, Υπουργείου Εξωτερικών. Έχετε όμως πολλούς, πολλούς περισσότερους από τον υπαλλήλου και έχετε μάλιστα και πάρα πολλά αυτοκίνητα που έχετε παραγγείλει. Κλείνουν οι πρεσβείες σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και οι Βρετανοί είναι αναγκασμένοι ε, να ταξιδεύουν όλο και περισσότερο ε, το World ε, της BBC και αυτό υφίσταται περικοπές. Ε, θέλω λοιπόν σε έτσι δύο πράγματα. Μήπως μπορούμε να έχουμε πίσω τα λεφτά μας, γιατί εμείς μπορούμε να τα δαπανίσουμε καλύτερα, να τα ξοδέψουμε καλύτερα. Και δεύτερον, επειδή αυτή η υπηρεσία δεν ε, έχει κερδίσει εξοπιστία ούτε για την Αίγυπτο, ούτε για τη Λιβύη, τότε τι νόημα έχει να εξακολουθήσει να υφίσταται η υπηρεσία αυτή. La parola το λόγο έχει η Βαρόνη Άστο να την ακούσουμε με προσοχή. Ωραία, ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση που μου θέσατε είναι τι, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα αυταρχικά καθεστώτα και αν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε την διαδικασία που ακολουθούμε. Το έχω ήδη πει και νομίζω πως κάτι που προκύπτει από αυτόν τον γύρο των συζητήσεων είναι αυτό το θέμα του πότε και πώς συμμετέχουμε και πώς εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τη συμμετοχή μας ώστε να απομακρυνθούμε όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ε, υπάρχουν διάφορα που μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε την ισχύ αυτής της Ένωσης στα μάτια των τρίτων χωρών. Είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς πώς κάθε λέξη που λέμε, οι δηλώσεις που εμείς κάνουμε και εγώ κάνω, ε, α, τις διαβάζουν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σχολιάζονται από εκείνους που προσπαθούν να αλλάξουν τα καθεστώτα. Έπειτα η δυνατότητα δυνατότητα οικονομικών κυρώσεων που χρησιμοποιούμε με στόχο άτομα ε, ή καθεστώτα ε, επίσης ε, ασκούν τεράστια πίεση. Παραμένω στην αρχή ότι εκεί που μπορούμε να συμμετέχουμε για να επιτύχουμε την αλλαγή και θα πρέπει να έχουμε ένα φάσμα ανάμεσα στην απομόνωση και την πλήρη συμμετοχή για να μπορούμε να κινηθούμε. Και ένα από τα πράγματα, που, τα νέα στοιχεία μάλλον στην ε, πολιτική κοινωνία είναι ακριβώ να μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό πιο σωστά. Κυρία Δεκαζέρα, για την Ιαπωνία, εγώ νομίζω ότι καλά τα πήγαμε όσον αφορά τη στήριξη που προσφέραμε αμέσω στην Ιαπωνία. Ξέρετε ότι μας ζήτησαν ε, βοήθεια, ε, την προσφέραμε, δεν τη χρειάστηκαν στη συγκεκριμένη στιγμή και μετά επισήμως μας ζήτησαν βοήθεια και το κάναμε. Ε, και θα είναι συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων. Καταρχήν χρειάζονται στήριξη που να μπορεί να σταθεί από μόνη της στο επιτόπου, γιατί στις πιο ε, πληγεί στι περιοχές ε, πρέπει να μπορούμε να φτάσουμε και να μείνουμε εκεί, δηλαδή με τη γλώσσα να μιλάνε, ε, τρόφιμα να μπορούν να δώσουν όσον αφορά το συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και αυτό βαραίνει την περιτροπή προεδρία και πρέπει να επενέσουμε την Ουγγαρία που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Οι πρέσβεις επιτόπου τα κατάφεραν μια χαρά. Μπορούμε να πάμε καλύτερα. Ναι, μπορούμε και καθημερινά αυτό το εξετάζουμε, αλλά θα πρέπει όντω να είναι πιο σωστό ο συντονισμό μα. Κάνουμε πολλά είδη στι Βρυξέλλε γιατί μπορέσαμε να στηρίξουμε την Προεδρία και να γίνει σωστό συντονισμό, αλλά σίγουρα στην αρχή είναι δύσκολο να επιτευχθεί και έχετε δίκιο που το θίγετε για το Σουδάν. Όπω ξέρετε, έχουμε μια νέα στρατηγική που προσπαθεί να βασιστεί στην αναπτυξιακή βοήθεια, την πρόληψη των συγκρούσεων και νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα που είναι θαρρυντικό ε, μάλλον που είναι η ενθάρρυνση και η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Σουδάν και επίση να υπάρξει ισορροπία με το Βόρα. Εγώ ανησυχώ για το τι συμβαίνει στον Ταρφούρ αυτή τη στιγμή, όπου η βία αναζωογονείται και μα ανησυχεί πολύ. Και προσπαθούμε ακριβώ να σκεφτούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε εκεί. Κύριε Πρέντα, προηγμένη κατάσταση και ο δικό χάρτη. Συμφωνώ και πάλι. Προσπαθούμε όντως να αναθεωρήσουμε την ε, πολιτική γετνήσεις με βάση τα μέσα που έχουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη με σημεία σε αυτόν τον χάρτη που θα μας ε, διευκολύνουν να δούμε πόσο αποτελεσματικοί είμαστε. Είμαστε. Ένα παράδειγμα επίκαιρο είναι ότι στην Αίγυπτο, συζητώντα με τον νέο ε, Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Συντονισμού, ε, ε, είδαμε ότι πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε και ταυτόχρονα το ίδιο και για τους υπόλοιπους. Η αμοιβαία δηλαδή ε, αποδόση λογαριασμών είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε χρήματα για να φτιάξουμε τη δημοκρατία. Πρέπει να δούμε και τη δημοκρατία να οικοδομείται. Αν λέμε ότι στηρίζουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι όντω εκεί πάντα λεφτά, ότι είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά να είμαστε και απαιτητικοί. Θέλουμε να έχει ο κόσμο την ευκαιρία να το κάνει αυτό και να έχει και του απαραίτητου πόρου για να το επιτύχει. Ναι, ε, πήγαμε στη Βενγάζη, το, αυτό που είδαμε, γιατί μιλήσαμε με διάφορες ομάδες επιτόπου, είδαμε κόσμο που είναι ξεκάθαροι και λένε ότι θέλουν δημοκρατία, θέλουν ελευθερία. Βρήκε επίσης ε, αρκετή αποφασιστικότητα στον κόσμο εκεί να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία ώστε να γίνουν οι αλλαγέ. Αυτό ήταν πριν βέβαια να ξεκινήσει ο πόλεμος, πριν να φτάσει ο κατάφη κοντά στη Βενγάζη. Υπήρχε δηλαδή μια νευρικότητα για το μέλλον. Επίσης έλεγξε να υπάρχουν αρκετοί πόροι. Τότε είχαν αρκετούς πόρους. Και ενώ συζητούσε με την ε, Ερυθρά η Μισελνο να δουν τι ακριβώς μπορούσαν να κάνουν, τώρα όμως πρέπει με πιο μακροπρόθεσμα να δούμε για να το στηρίξουμε όχι μόνο στα σύνορα αλλά και αλλού. Καθώς ελπίζουμε ότι θα αρχίσουν να πορεύονται προς τη δημοκρατία. Πολύ χρήσιμη επίσκεψη και πολλές πληροφορίες. Είναι μια σύντομη υπερώτηση. Όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα του Εθνικού Μεταβατικού Συμβούλου, κάνετε κάποια αξιολόγηση. Από όσο γνωρίζουμε, το Συμβούλιο αποτελείται από 31 ανθρώπους. Ορισμένοι προέρχονται από το καθεστώς ε, άλλοι όχι, άλλοι εκτός της Λιβύης, άλλοι εκτός. Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω κρίση, ε, απλώς ε, πρόκειται για ένα σημαντικό συνομιλητή και αλλά ο λαός θα αποφασίσει ποιο θα, ποιος θα είναι ο του και σίγουρα θα συζητούμε μαζί τους. Επίσης γνωρίζετε... Ο Ρόμπερτ δεν μου έδωσε πληροφορίες για τους ε, διάφορους ε, υπουργούς. Σίγουρα ορισμένοι ε, Βρετανοί στο κόμμα σας ε, θα εξοργίζονταν να πρότεινα επιπλέον ε, πόρους για καμιά δεκαριά υπουργούς όπως είπατε. Τώρα ξέρετε πόσο μου είναι το θέμα της Γάζας ε, και πόσο έχω προσπαθήσει να υπάρξει πρόσβαση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες στη λωρίδα της Γάζας για να αναπτυχθεί η οικονομία και πόσο σημαντικό θεωρώ ότι είναι αυτό. Και επίσης ανησυχώ για τις ε, επιθέσεις ε, πυράβλων που προέρχονται από τη Γάζα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε το άνοιγμα και έχουμε προτείνει 5,5 εκατομμύρια που έχουμε ώστε να βελτιώσουμε τις υποδομές και να ανοίξει όντως ε, ε, το σημείο διάβασης, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα, ώστε ο κόσμος μέσα στη Γάζα να αισθανθεί πως έχει ευκαιρία, έχει μέλλον, ιδιαίτερα οι νέοι. Κύριε Παντζέρη τώρα, η Αφρικανική Ένωση, ναι, πολύ σημαντική, συναντώνται την Παρασκευή, εγώ είχα επαφή μαζί τους και φυσικά η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική εταίροι μαζί μας. Κυρία Χάουταλα, για τη Συρία, ναι, ανησυχώ και εγώ για το τι συμβαίνει. Παρακολουθούμε ότι εκεί υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις βίας στις πόλεις και πάλι ε, το θέμα της ε, συμμετοχής ή της απομόνωσης και ήδη είχαμε κάποια μηνύματα. Πρέπει να παρακολουθούμε τις επόμενες ώρες τι συμβαίνει. τα Citizen είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων, δηλαδή πληροφόρηση πολύ γρήγορα για το τι συμβαίνει επί τόπου ε, ενημέρωση ταυτόχρονη δηλαδή, Και επίση συγκέντρωση πληροφοριών που μπορεί να μας βοηθήσει για να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις ε, Αν έχετε άλλες ιδέες ευχαρίστω να μας τις δώσετε. Κύριε Μάντλενερ, διαφωνώ μαζί σας Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα άλλο. Από τη μια μου λέτε ότι είμαι άχρηστη, από την άλλη με ρωτάτε τι κάνω για όλα αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ ότι εμένα είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση, δεν συμφωνώ με τη δική σας ανάλυση όμως και νομίζω πως η συνάντηση με τον Εξυπουργό Εξωτερικών, πράγμα που έκανα πρόσφατα, και ότι ε, όσα λέει ο Πρόεδρος, αλλά λέει και η αντιπολίτευση, είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τη χώρα αυτή, γιατί έχει πολύ πολύ βαθιά προβλήματα. Και ξέρω πως δεν συμφωνείτε μαζί μου ή με το τι κάνει η υπηρεσία μου, αλλά ο σεβασμός που τη χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ολλανδοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολόκληρο τον κόσμο, μην το υποτιμάτε αυτό. Πολλοί, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι τα όσα κάνουμε είναι καταπληκτικά. Προσπαθούμε να το στηρίξουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και είναι δική μου, δικό μου προνόμιο το να μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Κάθε πέντε χρόνια ε, ναι, αλλάζω αυτοκίνητο, αλλά αυτό γινόταν ε, και στα άλλα, σε άλλες, άλλες υπηρεσίες όπου εγώ υπηρέτησα. Ε, εντάξει, μπορείτε να λέτε, να βγάζετε διάφορα από τα άρθρα, να μιλάτε για χιλιάδες αυτοκίνητα, μα εσείς τα ξέρετε καλύτερα, περίμενω καλύτερες, ε, καλύτερα σχόλια. Οπότε κοιτάξτε να βρείτε τουλάχιστον τα σωστά στοιχεία. Εντάξει, ε, είστε απόλυτα ελεύθερος να έχετε αντιρρήσεις για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ότι μπορεί να θέλετε να έχουμε 27 εκπροσώπους και όταν ε, συναντώμεθα να έχουμε κάτι να πούμε. Εγώ νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από το τι κάνει ε, από μόνη της η Ολλανδία ή η Βρετανία. Αυτή η βρετανια Α, σχέση μεταξύ των κρατών είναι σημαντική και προσπαθώ με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και με το σεβασμό, όλο το σεβασμό στους φορολογούμενους Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνω ό,τι μπορώ και να γνωρίσουμε το δύσκολο έργο. Εάν όταν ο κόσμο αλλάζει τόσο πολύ και αν δεν επενδύσουμε στο μέλλον των λαών στην νότια γειτονιά μα, εμεί θα το πληρώσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και να το κάνουμε. Πρόεδρος, ε, τρίτος λοιπόν ε, γύρος ε, ερωτήσεων, συνάδελφος Λάντσπεργκη, σας υπενθυμίζω 1,5 λεπτό και δυνατόν μία μόνο ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε και αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτική μας απέναντι στη Λιβύη. Εσείς προσωπικά και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε παραλάβει ότι έχει χάσει κάθε νομιμότητα το καθεστώς του Καντάφη θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την πρωτοβουλία της Ρωσίας να διαμεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις και να επαναφέρει ένα τμήμα της νομιμότητας, νομιμοποίησης του Καντάφη που τον αναγνωρίζουν ως μέρος διαπραγμάτευσης σε μία σύγκρουση. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε περισσότερη πληροφόρηση, ε, ποια είναι η θέση για μια, ένα κράτος που δεν υποστήριξε ε, τα Ηνωμένα Έθνη και πώς διαπραγματεύονται στη Βενγάζη με κάποιο συμβούλιο που μπορεί να δημιουργήσει διχοτόμηση στη Λιβύη με στόχο που μπορεί κάποιοι να έχουν να έχουμε μια νέα μεγάλη παγωμένη σύγκρουση αυτή τη φορά στη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ κυρία Κοπά και ο ε, Κύριε Πρόεδρε, θα γυρίσω πάλι στη Λιβύη. Δεν ακούσαμε μια στρατηγική ανάλυση για το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή και για την ευρωπαϊκή θέση. Εδώ είχαμε ένα νοηματικό άλμα. Από την έναρξη του δημοκρατικού κινήματος περάσατε στην ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση και φυσικά στόχος είναι η προστασία των αμάχων Όπω και αργότερη η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου, πράγματα που όλοι συμφωνούμε. Η ερώτησή μου είναι ποιο είναι συγκεκριμένο ο στρατιωτικό στόχο μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φύγει ο Καντάφη, να διαπραγματευτεί με του εξεγερμένου και πώ το επιδιώκουμε. Υπάρχουν σήμερα διεύλοι επικοινωνίε με τον συνταγματάρχη Καντάφη. Δεύτερο ερώτημα. Τι έχετε σκοπό να κάνετε για να συντονιστούν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή η Ένωση δείχνει να συνθλίβεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τις πολιτικές των κρατών μελών. Και τρίτο σημείο, την προηγούμενη εβδομάδα στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, ο κύριος Ποπόφσκι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας είπε ότι η υπηρεσία σας προχωράει σε, όπως ο ίδιος είπε, prudent planification για την περίπτωση της Λιβύης, χωρίς όμως να μπορέσει να εξηγήσει στην Επιτροπή τι σημαίνει αυτό. Μπορείτε εσείς σήμερα να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Grazie, collega Watson. Όχι, ε, ο κύριο Αγκουράκης. λοιπόν. Ε, θα ήθελα να σα ε, συγχαρώ για τα επιτεύγματα. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να σα κάνω τρει ερωτήσει που και τρει έχουν σχέση με τη Λιβύη. Ε, πρότεινε εξή. Ε, υπάρχει η έκκληση του Αραβικού Συνδέσμου για απαγόρευση ζώνης ε, πτήσεων ε, και θα ήθελα να ρωτήσω. εσείς συνεργαστήκατε με τον Αραβικό Συνδεσμό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό συμφωνείτε μαζί του. Ο, ο κύριος Γκαντάφη βομβαρδίζει, συνεχίζει να βομβαρδίζει άμαχο πληθυσμό στη Μισράτα και αλλού και θεωρείται λοιπόν ότι ο Καντάφη μπορεί να αποτελέσει και αυτό στόχο, νόμιμο στόχο. Δεύτερη μου ερώτηση. Εχθές στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έγινε συζήτηση για το ποιος τελικά είναι ο στόχος της παρέμβασής μας και εσείς πώς περιγράφετε το στόχο αυτό της επέμβασης. Και το τρίτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, αν αποσυρθεί από την ηγετική θέση, πιστεύετε ότι θα πρέπει να λάβει το ΝΑΤΟ ή ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αγκουράκης και μετά κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Αραβικός Σύνδεσμος από ό,τι μαθαίνουμε έχει αποσύρει την υποστήριξή του στην επιχείρηση την, ε, στον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο ενάντια στη Λιβύη. Το θέμα είναι, η κύριε Άστον, τι γνώμη έχει εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι ε, της απόφασης ε, του Συμβουλίου στις, ε, στις 11 του Μάρτη, η οποία, οι οποίοι όροι ήταν ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που το ΝΑΤΟ είχε αποφασίσει στις 10 του Μάρτη όσον αφορά την επέμβαση στην Λιβύη. Τα λέω αυτά, κυρία εκπρόσωπε, γιατί έχω τη γνώμη ότι αυτός ο πόλεμος είναι εντελώς παράνομος, είναι εντελώς παράνομος και με όρους του Ιμανουήλ Καντ από ό,τι λέει ε, η μεγάλη γερμανική εφημερίδα. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να τελειώσει εδώ και τώρα ε, αυτός ο ανελέητος ε, βομβαρδισμός. Πρέπει να τελειώσει γιατί είναι ένας συμπεριαλιστικός πόλεμος ο οποίος δεν έχει να κάνει ε, σε τίποτα με την παραβίαση ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων που πραγματικά το καθεστώς Καντάφη έχει κάνει. Εξάλλου ο γιος του, όπως ξέρετε, έχει κάνει διατριβή στο Oxford και έχει σπουδάσει στην Αυστρία και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχουμε παρόμοιες καταστάσεις και στο Μπαχρέιν και στην Γεμένη αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν βομβαρδισμοί και καλώς δεν φαντάζομαι τώρα τα βρετανικά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν ε, τη Γεμένη και ξέρω εγώ κάποια άλλοι ε, ε, τον Μπαχρέιν. Τέλος, ε, θέλω να τοποθετηθείτε σε δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Βελγίου του Υπουργού Στρατιωτικών του Βελγίου, ε, ο οποίος χθες δήλωσε ότι βεβαίως υπάρχει ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη, στη Λιβύη, που για μένα ακριβώς αυτό θα γίνει. Και θα έπρεπε να είμαστε πιο ειλικρινεί κύριε Άστον, να μας πείτε αυτά που ξέρετε, ότι δηλαδή θα υπάρχει κατοχή στη Λιβύη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. La parola al collega το συνάδελφο κύριο Βανόρτεν και θα ακολουθήσει Βανόρτεν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, έχει έρθει η χρονική στιγμή για αλληλεγγύη και δεν είναι η στιγμή ε, για να επιδιώξει κανεί τι φιλοδοξίε των ευρωπαϊκών θεσμών και βεβαίω η ΚΕΠΑ μπορεί να μην έχει σημασία αλλά ίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει με άλλου τρόπου και εγώ προτείνω τρει συγκεκριμένα. Πρώτον, να ε, επιβεβαιώσει την Τουρκία ότι έχει θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να τη στηρίξει, δεύτερον να ενθαρρύνει την ε, στράτευση των Αράβων και τρίτον οικονομική βοήθεια έχοντας κατά νου ότι λείπουν τα χρήματα. Θέλω λοιπόν κύριε Πρόεδρε να πω ότι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη συνεισφέρει κατά, με 16 δις ε, στην, συνεισέφερε τελευταία 15 χρόνια στην οικονομία των χωρών της Βορείου Αφρικής και ρωτώ την κυρία Άστον τι ακριβώς θα κάνετε για να αλλάξετε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί φαίνεται ότι τα χρήματά μα δεν έπιασαν τόπο. Πώς μπορείτε λοιπόν να αλλάξετε την κατάσταση. Αναφέρατε πόσο απασχολημένοι ε, είσαστε, εγώ θα έλεγα να περιορίσετε ίσως τα ενδιαφέροντά σας και να εστιάσετε την προσοχή σα σε ένα δύο. Και όσον αφορά το θέμα των χρημάτων, Α ξεχάσουμε τα αυτοκίνητα, αλλά τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ που εδόθησαν ε, σε διαγωνισμό ε, για ε, δημόσιες σχέσεις και προαγωγή των δημόσιων σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, Χάις Ντόφλα και επόμενος Γκάλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν έχουμε επαναστατικές ε, δράσεις, αυτές έχουν το δυσάριστο ότι σε μεγάλο βαθμό παραμένουν ε, κάτω, εκτός ελέγχου και στη τελική ανάλυση αυτό το οποίο προκύπτει είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι. Από ό,τι φαίνεται όμως, οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή ε, έχουν ξεφύγει εκτός ελέγχου και έτσι κύριε Λάμπστορφ ε, αυτά που λέει ο κύριος ε, Μπέστεμπελε που είναι απλά προσευχές δεν είναι και πολύ καλύτερα ε, είπε το τι ακριβώς είναι απαραίτητο για να έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, όμως τα πράγματα δεν λειτουργούν τόσο απλά. Και έχω μία ερώτηση προς εσάς κυρία Ήπατη εκπρόσωπο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Μπαχρέιν στο μέλλον. Το γεγονός ε, ότι ε, συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μια πλατεία, κατασφαγιάζονται. Αυτό μας θυμίζει την Κίνα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι μπροστά από τον Μπαχρέιν είναι ο Αμερικανικός στόλος και κάτι άλλο. Ε, γιατί χτίσαν πολλά εδώ. Το ωραίο σε ένα δημοκρατικό σύστημα είναι ότι ακόμα κι αν πονάει κάτι, ακούει κανείς βλακίες, αλλά ε, παρόλα αυτά, ακόμα κι αν υπάρχουν ε, πολιτικά τυφλοί, ε, δυστυχώς είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό οφείλεται σε κάποιους συναδέλφους. συνάδελφος Γκάλ και επόμενος Κέλαμ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στη Λιβύη, εσείς αναφερθήκατε ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια γύρω ε, και μέσα στη Βεγγάζη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αναπτύσσει δραστηριότητε και ρωτώ, χρειαζόμαστε ανθρωπιστική αποστολή και επιχείρηση μέσα στη Λιβύη και ίσως ε, χρειαζόμαστε και να την προστατεύσουμε με στρατιωτικά μέσα. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά την Ουκρανία, είπατε θα πάτε εκεί σύντομα και σας ε, καλώ να μην εστιάσετε τη συζητή σας μόνο στην ζώνη ελεύθερων πολιτικών ανταλλαγών, αλλά παρακαλώ να επισημάνετε το ότι υπερίζεται όλο και περισσότερο η δημοκρατική θεσμή και παρεμφανίζεται η εξουσία της Ρωσίας σε όλα τα επίπεδα. Τέτοιου είδους λοιπόν Συμπεριφορέ. συμπεριφορές νομίζω ότι δεν μπορούν να ε, οδηγούν σε στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος και μετά η κυρία Γκόμης. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, πριν δύο εβδομάδες το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε συνεπή εξωτερική πολιτική σαφώς υπέρ των ε, δημοκρατικών δυνάμεων. Κάνετε πολύ καλή δουλειά τον ε, τελευταίο καιρό και συμφωνώ πως δεν είναι θέμα συντονισμού, πρόκειται για διαφορετικές απόψεις ε, των ε, ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ωστόσο, μπορώ να σας ρωτήσω, μπορούμε να αποκομίσουμε διδάγματα από την κρίση του, της Βόρειας Αφρικής. Η σημερινή πολιτική είναι πιο πρακτική και ρελαστική από ό,τι παλιότερα, δεδομένη της εντυπωσιακή ζήτηση για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Και έπειτα, θα ήσασταν έτοιμοι να σχεδιάσετε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για όλα τα αυταρχικά καθεστώτα. Όπως είπε και ο κύριος Μπράντερ, χρειάζεται μια δραστήρια εξωτερική πολιτική, όχι μόνο να τη δράμε κατόπιν ορθής. Και έπειτα, εφόσον αυτή η αλλαγή υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου έχει καταστεί δυνατή με πολύ αναπάντεχες ε, καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να μην μείνει μόνο στις ε, θεωρίες αλλά να περάσει σε realpolitik. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε δίνοντας το λόγο για 10 λεπτά στην ύπατη πρόσωπο. No, Gomez, scusa. Και το μόλι τα σκούζα, αλλά κολέγγα εγώ. Α, ζητώ συγγνώμη από τη συνάδελφο Γκόμε. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω και εγώ την επαφή μαζί σα μέσω του κ. Βημόντα για την Βόρεια Αφρική και θα ήθελα να πω πω λυπούμε γιατί η ΚΕΠΑ δεν κινητοποιήθηκε για το σχεδιασμό και το συντονισμό για την εφαρμογή της ε, ζώνης απαγόρευσης πτήσης, αλλά μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους. Μπορεί να πείτε αν τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν. Αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να μην σας ε, έδωσε την ομοφωνία, αλλά σίγουρα σας έδωσε την δυνατότητα να αναλάβετε πρωτοβουλία και να θέσετε τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις. Τώρα συμφωνώ πόσο φρικτή είναι αυτή η απόφαση για τη δήλωση για τους διαδηλατές, για τον Μπαχρέιν. Συμφωνώ και εγώ. Ανησυχώ πολύ γιατί δεν υπήρξε ε, καμιά αναφορά στην παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας στην καταστολή. Έστειλαν εκεί στρατεύματα για να καταστήλουν το λαό του Μπαχρέιν. Και αυτό δεν μας δίνει αξιοπιστία στον αραβικό κόσμο. Καταλαβαίνω τώρα το ρόλο και το νόημα του νέου σχεδίου Μάρσαλ, τα τρία αρχές για τι οποίε μιλήσατε, αλλά και εγώ έρχομαι χτε από την Αίγυπτο, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολύ καλή εικόνα, ε, γιατί ακριβώ η αντίληψη είναι ότι στηρίξαμε τον Μουμπάραγκ μέχρι τέλους. Υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα για το λαό που πρέπει εμείς να στηρίξουμε, η δημοκρατία, κρατός δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, η κατάσταση των γυναικών και χρειάζεται διπλωματία και για αυτά τα θέματα. Τώρα έχετε το λόγο για 10 λεπτά, στα αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαντσμπέρκης, ρωτήσατε για τη χαμένη νομιμότητα του Γκαντάφη και την πρωτοβουλία της Ρωσίας, την οποία δεν γνωρίζω. Δεν έχω ε, καταλάβει ακριβώς ποια θα ήταν αυτή η πρωτοβουλία των Ρώσων. Αλλά εμείς θεωρούμε σίγουρα ότι ο Καντάφη έχει χάσει την νομιμότητα και ότι οποιαδήποτε ε, έκβαση θα είναι η δυνατότητα του λαού να ε, έχει νέα ηγεσία. Δεν θέλουμε καθόλου ε, παγωμένη σύγκρουση εκεί. Θέλουμε μια χώρα με εγγυημένη την ε, δαφική της ακαιρεότητα. Άλλωστε αυτό είναι και τμήμα του ψηφίσματος. Η κυρία Κοπά ρώτησε για διάβλους επικοινωνίας και ότι συνθλίβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στους διάφορους οργανισμούς, κυρία Κοπά. Ε, το prudent planning, η σόφρον ε, πολιτική προγραμματισμού και σχεδιασμού ήταν ε, ότι διερευνήσαμε μία σειρά δυνατοτήτων δεν καθυστερήσαμε να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει ε, αμέσω, αλλά ε, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού εξετάσαμε διάφορα ενδεχόμενα για την αυτιλιακή υποστήριξη, για παράδειγμα, ή την υποστήριξη για καποιου που θέλουν να φύγουν από τη ε, Λιβύη και χρειάζονται υποστήριξη θαλάσσια. Άλλοι εξέτασαν, όπως και το ΝΑΤΟ, ε, την ε, θαλάσσια επιτήρηση του εμπάργου των όπλων. Ή επίσης ε, τι γίνεται με εκείνους που μπαίνουν στη Λιβύη από τα νότια σύνορα της. Υπήρχαν διάφορα ενδεχόμενα. Επίσης εκένωση του πληθυσμού εκεί σε μεγάλο βαθμό, τι γίνεται στα σύνορα, πώς επαναπατρίζονται άνθρωποι που δεν είναι ε, κάτοχοι ευρωπαϊκών διαβατηρίων, δεν είναι πολίτες της Ένωσης, τι θα γίνει με τους Αιγυπτίους που είναι στα τινησιακά σύνορα κτλ. Ε, ε, δηλαδή υπάρχουν διάφορες δυνατότητες που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να τα κάνει αυτά και μεταξύ αυτών και στρατιωτικά μέσα. Από το σχεδιασμό μετά λοιπόν περνάμε στις αποφάσεις όπου 27 κράτη αποφασίζουν τι πρέπει να γίνει. Κάθε χώρα είναι κυρίαρχη για αυτά τα θέματα. Εμείς κάνουμε το σχεδιασμό και το συντονισμό, αλλά τα κράτη-μέλη αποφασίζουν και έρχονται μετά στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τα θέματα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαστε ε, φρόνιμοι ακριβώ γιατί είμαστε και προσεκτικοί στη δράση μα. Ο κύριο Γότσον. Όχι ερωτήσει, ο πρόεδρο, δεν μπορώ να δεχτώ. Για την επικοινωνία. Με του διάβολου επικοινωνία τι εννοείται, με τη Λιβύη. Α, είχα σημειώσει, ναι, αυτό το διάβολο επικοινωνία. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άμεση ε, υπάρχουν εκπρόσωποι του καθεστώτος ε, και γνωρίζω ότι ταξιδεύουν ε, εντατικά και προς τα Ηνωμένα Έθνη. Το θέμα είναι πώς θα συνεργαστούμε με τους πολίτες, με το λαό για να έχει το μέλλον που θέλει. Αυτό είναι το σημαντικότερη πρόκληση. Λοιπόν, Βότσον, τρεις ερωτήσεις. Ζώνη απαγόρευση ο αραβικός σύνδεσμος. Είχαμε επαφή μαζί του. Σήμερα μίλησα με τον Άμρ Μούσα είναι καλή σχέση μας, είχαμε από την αρχή ε, της ανάληψης των καθηκόντων μου ε, συχνές ε, τακτικές συναντήσεις και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά ε, για το θέμα του μέλλοντος, γιατί αναγνωρίζω ε, ότι βέβαια θα φύγει από τον Αραβικό Σύνδεσμο γιατί θα είναι ε, υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο με το διάδοχό του. Συνεργαστούμε πάρα πολύ γιατί είναι τεράστια σημασία ε, αυτής της συνεργασίας και στόχος μας. Ερωτήσατε τώρα ποιος είναι ο απότερος στόχος. Στόχος είναι να μπορέσει ο λαός της Λιβύης δημοκρατικά να επιλέγει την κυβέρνηση που θέλει. Ε, είχαμε ε, συναντήσεις, συνεννοήσεις με Λιβύους και εκτός και εντός της Λιβύης. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη φιλοδοξία τους και αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να τους επιτρέψουμε να το πράξουν αυτό. Είναι σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράδοση της διοίκηση από τις Ηνωμένε Πολιτείες το συζητάνε με το ΝΑΤΟ. Αυτό τον καιρό κάνει το σχεδιασμό το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εκείνοι θα το αποφασίσουν. Αλλά συζητήσεις με το ΝΑΤΟ ε, μάλλον ε, δείχνουν ότι προς τα εκεί θα κατευθυνθούμε. Κύριο Αγκουράκη, είπατε ότι οι όροι τη 11 Μαρτίου ήταν οι ίδιοι με τη 10η Μαρτίου ε, ήμουν εγώ σε εκείνη τη συνεδρία δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι παράνομο ε, δίνει νομιμότητα το Συμβούλιο ασφαλεία και απόφαση του το ψήφισμα 1973 οι όροι και οι προποθέσει είναι σαφείς ε, πληρώθηκαν και ανανελήφθη δράση σέβομαι το δικαίωμα κάθε χώρας να κάνει ό,τι πιστεύει ε, πέρασε το ψήφισμα χωρίς καμία ψήφο κατά και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Βανόρντεν, για την Τουρκία, συμφωνώ απολύτως, είναι πραγματικά κρίσιμος εταίρος και θέλω να συμμετέχει η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκαθεν το πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω γιατί η συνεργασία με την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο με τους ε, Τούρκους στη συνεργασία γιατί διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο. Επίσης, το θέμα της δέσμευσης των αραβικών κρατών είναι τεράστια σημασία για μα, και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τα χρήματά μας, να πιάσουν τόπο. Δεν δέχομαι ότι όλα τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει πήγαν χαμένα. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά. Ε, μιλούμε με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών που λένε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Μα αυτό είναι καλό σημάδι ότι κάτι έχουμε κάνει και είναι πολύτιμη οικονομική συνεργασία. Δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάντα θα πρέπει να προσπαθούμε. Αυτό είναι απόλυτη προπόθεση. Βεβαίω είναι σε τελική ανάλυση χρήματα των φορολογουμένων και θα πρέπει να είναι προ όφελο και των λαών τη Ευρώπη να δουν εκεί τη σταθερότητα και τι πραγματικές ευκαιρίες ε, και εμπόριο. Είναι καλό αυτό. Και το 8,6 εκατομμύριο που με ρωτήσατε είναι πενταετές πλαίσιο και σύμβαση για το σύνολο ε, της εξωτερικής ε, δράσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλο τμήμα υποστηρίζει το Euronews στα φαρσί, στα περσικά και είναι μεγάλη προσπάθεια και μέλημα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό. Και ε, βεβαίω δεν είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ε, αυτό εμπέπτει λίγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για τη σύμβαση αυτή, αλλά είναι πενταετή για να βεβαιωθούμε ότι θα μπορούμε να ε, δημοσιοποιούμε τη δράση μας και να έχουν οι αντιπροσωπείες υλικό για να μπορούν να, να προβάλλουν την Ευρώπη. Για το Μπαχρέιν, το Σαββατοκύριακο Είχα στείλει ε, ένα απεσταλμένο στο Μπαχρέιν. Δύο φορές συναντήθηκα με αποστολή, αντιπροσωπεία ε, του βασιλέως και πήγε στη Σαουδική Αραβία. Ε, τα πράγματα θα πρέπει να ηρεμήσουν. Ρώτησε ο κύριος Λάμστροφ τι γίνεται με τα συμπεράσματα για τον Μπαχρέιν. Νομίζω ότι είναι δίκαια. Το ξανακοίταξα, είναι ισορροπημένο. μήπως είχα ξεχάσει τίποτα. Ε, μιλούμε για το ρόλο των κρατικών αρχών των υπηρεσιών, ε, καλούμε ε, όλους σε συγκράτηση και σε ηρεμία. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε το διάλογο, χωρίς προαπαιτούμενα, πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να γίνει. Ο Ρόμπερτ Κούπερ τώρα εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή και σε τελική ανάλυση η δουλειά μας είναι να προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τις συγκρούσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Γκάλερ, Λιβύη και την πολιτική αποστολή. Η προστασία των στρατιωτικών. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε τι διαθέτουμε, τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Σας είπα προηγουμένως, η κένωση του πληθυσμού χρειάζεται καμιά φορά και στρατιωτική υποστήριξη. Να γίνεται σωστή η εκμετάλλευση των μέσων, αλλά χωρίς σύγχυση. Όταν κάνουμε πολιτικές αποστολές με βοήθεια προς τον πληθυσμό είναι τελείως διαχωρισμένο από την οποιαδήποτε ε, στρατιωτική επέμβαση. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους. Και συμφωνώ για την Ουκρανία. Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι θα προχωρήσουν ε, στις δημοκρατικές ελευθερίες. Στο θέμα της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου έχω απογοητευτεί γιατί δεν προχωράει πιο γρήγορα γιατί και εκείνοι δεν προχωρούν γιατί είναι προς όφελος χώρες. Κύριε Κέλαμ, ε, προληπτική ενεργή πολιτική. Ε, ορισμένα από αυτά που λέω και γράφω σε άρθρα μου ε, έχουν να κάνουν με το πώς θα προχωρήσουμε. Σας λέω ότι δεν είναι τα πιο προβεβλημένα, τα πιο ένδοξα, αλλά είναι τα πιο σημαντικά αυτά που κάνουμε. Και η προληπτική δράση είναι ότι συζητούμε με ε, χώρες. Η Ορδανία, έχω αποστολή αυτή τη στιγμή στην Ιορδανία. Συζητούμε για μεταρρυθμίσεις πολιτικές. Έχουμε στείλει επεσταλμένους στον Μπαχρέι να συζητούν. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τις χώρες γιατί θέλουμε να βλέπουμε τη δημοκρατία και την ελευθερία, αλλά όχι το χάος. Να μπορεί ο κόσμος όσο γίνεται απρόσκοπτα να μεταβαίνει στη δημοκρατία. Και τέλος για την κυρία Γκόμες. Δεν συμφωνώ με την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Αίγυπτο. Έχω πάει δύο φορές ε, Είμαι διατεθειμένη να δεχτώ τις επικρίσεις ε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει, και είστε και πολύ ευθεία μαζί μου, έχετε δίκιο. Και είναι γεγονός αυτό. Αλλά ε, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι προσπαθούν με γνήσιο τρόπο, με ειλικρινή, να ε, προχωρήσουν και εμείς να είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε. Και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διδραματίσει το ρόλο της εκεί, αλλά περισσότερο από τίποτα άλλο οι χώρες αυτές ανήκουν στους λαούς τους και οι λαοί θα αποφασίσουν το μέλλον τους, εμείς θα τους βοηθήσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταίος γύρος. Το λόγο έχει ο αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρούτσεκ και στη συνέχεια ο συνάδελφο Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο ε, Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Δεν πρέπει να έχουμε μια στρατηγική όσον αφορά αυτές τις χώρες. Όταν μιλάμε ε, για την ε, πολιτική νότου για τον ανάγκη διαθέτησης χρημάτων, όμως για τις χώρες του κόλπου εκεί δεν χρειαζόμαστε ε, να διαθέσουμε κονδύλια. Εκείνο που δεν κάνουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ άλλου είδου επαφέ, όμω εκείνο που δεν κάνουμε είναι να στηρίζουμε τη δημοκρατία. Και όπω πολύ σωστά είπατε, Χρειαζόμαστε τη δημοκρατία γιατί τελειώ δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα. Άρα δηλαδή μήπως ε, θα έπρεπε να αποφασίσουμε από κοινού με το Συμβούλιο Συνεργασίας ε, του Κόλπου μια στρατηγική όπου βέβαια θα διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας ε, στρατηγικής, επιχειρηματικά συμφέροντα όμως σιγά σιγά από κοινού με το Συμβούλιο αυτό να προχωρήσουμε προς το δρόμο της δημοκρατίας της ελευθερίας. Και η δεύτερη ερώτησή μου σε σχέση με την πρώτη μπορούμε να συνεργαστούμε ε, στο πλαίσιο αυτό και με την Τουρκία. Η Τουρκία αναφέρθηκε ήδη. Η Τουρκία ασκεί στην περιοχή και μεγάλη επιρροή γνωρίζει την περιοχή πολύ καλά. Ε, μήπως λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε και με την Τουρκία όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Κούκαν και μετά Αρλάκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βαρόνη, για το όσα μας είπατε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε να συζητήσετε μαζί μας και να μας ακούσετε. Η ερώτησή μου είναι συνέχεια συνέχεια των όσων είπε η κυρία Λούνατσα και το Κωσυφοπαίδιο. Περιμένουμε ακόμα να μας απαντήσετε. Θα έλεγα λοιπόν ότι το γεγονός ότι ο διάλογος Βελιγραδίου Βελιγραδίου-Πριστίνα ξεκίνησε είναι αν όχι επιτυχία σίγουρα είναι θετικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημά μου είναι, τι πιστεύετε εσεί για το μέλλον αυτών των διαπραγματεύσεων, γιατί διάβασα ότι πέρα από την αρχική καναμενόμενη συμμετοχή υπήρχε και ένας προσκεκλημένος από το State Department. Αυτό είναι όντω αλήθεια, θα καλέσετε και άλλου. Γιατί νομίζω ότι ο ένας που είναι εκεί ήδη αρκεί και περισσεύει. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν για τις εξελίξεις ή αυτές τις διαπραγματεύσεις και δεύτερο μου ερώτημα. Ποια είναι η κατάσταση και τι πιστεύετε εσείς για την έναρξη του διαλόγου με τις αρχές ε, του Κωσυφοπεδίου για τη διευκόλυνση θεωρήσεων για τον, τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σαρλάκη και επόμενη η παρέμβαση ο συνάδελφος Σάρκη. Ευχαριστώ κυρία Άστον. Δύο θέματα θέλω να σας αναφέρω και να ζητήσω τη γνώμη σας. Για εναλλακτικού τρόπους παρέμβασης στην τρέχουσα κρίση Μέση Ανατολής και ε, Βόρειας Αφρικής. Το ένα σχέδιο Μάρσαλ, καλή ιδέα. Ε, πρόκειται για μεγάλα ποσά, 10 δις σε 10 χρόνια. Σε τόσες πολλές χώρες ορισμένες είναι ήδη πλούσιες. Δεν νομίζω πως ε, θα είναι κάτι που θα έχει πραγματικά μεγάλο αντίκτυπο. Γιατί να μην εξετάσουμε άλλους τρόπους για να αντλήσουμε νέους τοπικούς πόρους που είναι πολύ ισχυροί. Πρώτος είναι το θέμα των, της ε, κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων που συγκεντρώνονται στο εξωτερικό από τους διάφορους τυράννους και τα δίκτυά τους, αλλά γίνει αυτό αυτό είναι ήδη ένα θέμα ε, επιτάπητος, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πολυμερές ε, μέτρο. Γιατί, μέσο, γιατί αν τα αφήσει στο κάθε, στο κάθε δεν πας πουθενά και, ή προχωράς πολύ αργά. Δεύτερο που μπορεί να αντλήσει ακόμα μεγαλύτερα ποσά είναι οι εξοπλισμοί στο περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Μιλάμε για τις πιο οχυρωμένες, τις πιο εξοπλισμένες χώρες στον κόσμο. 50 δις φέτος οι διαστρατικές δαπάνες συγκεντρωμένες στα 3, σε 3, 4, 5 άντε χώρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούσαν, να χρησιμοποιούσαν αυτούς τους εξοπλισμούς με λάθος τρόπο. Γιατί δεν μιλάμε για 50% περικοπή των εξοπλισμών και να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά να μπουν σε ένα ταμείο που θα είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη της περιοχής. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η συνάδελφος Σάρκη και μετά η κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Εμείς εκτιμούμε τις ε, διάκοπες προσπάθειές σας ε, να ακολουθήσετε τους ρυθμούς των αλλαγών και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με την κατάλληλη και ταχεία δράση. Για το Ιράν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ακολουθήσατε τα ε, αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά κυρίως του Ιρανικού λαού και λάβατε την απόφαση να επιβάλλετε επικυρώσεις σε ατομικούς παραβιαστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να ξέρω πότε θα έχουμε τον αντίστοιχο κατάλογο και πώς αξιολογείται το ρόλο του Ιράν στην περιοχή δεδομένης της ε, μεγάλης αναταραχής, κυρίως απέναντι στο Μπαχρέιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Νίπλερ και παρεμπόμενο θα είναι η Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Εδώ, εδώ κάθομαι. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ορισμένοι συνάδελφοι ήδη έτυξαν το Μπαχρέιν και την πολιτική στην Αραβική Χερσόνησο. Ε, ο συνάδελφος Κράτσερ Τόλφρε, η συνάδελφος, σας ρώτησε ποια είναι η πολιτική μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, σε ένα στόχο, σε ένα αποτέλεσμα στο Μπαχρέιν. Εσείς λοιπόν είπατε ότι μιλήσατε με τον Βασιλιά και μιλήσατε και με δύο υπουργού. Ε, λυπάμαι, αυτό δεν μπορεί να είναι σωστή απάντηση, μα δεν αρκεί. Και σα παρακαλώ πάρα πολύ, όπω και άλλοι συνάδελφοι εδώ το έκαναν, να ε, διατυπώνεται μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική και μια στρατηγική η οποία επιδιώκει στόχους και για το σύνολο της περιοχής ε, κύριε Αντιπρόεδρε δεν πρόκειται μόνο για το Μπαχρέν πρόκειται και για την Ιεμένη και ανησυχώ πάρα πολύ βλέποντας ότι μετά από παράκληση της ε, κυβέρνησης του Μπαχρέν επενεύει η Σαουδική Αραβία με στρατεύματά της. Ε, γι' αυτό λοιπόν σας ε, ερωτώ, θα κάνετε μια εντελεχέστερη ανάλυση. Τι θα κάνετε με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να κλείσει το θέμα με μια κουβέντα με τον Βασιλιά και δύο υπουργό. Πρέπει να κάνετε πιο διεξοδική έρευνα και συζήτηση. Και κάτι άλλο. Στη Λιβύη υπάρχει πόλεμος ε, από το Σαββατοκύριακο και εμείς ε, εδώ ε, συζητάμε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μα δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Ε, σας παρακαλώ ε, να αναλάβετε τον ηγετικό ρόλο και να μην περιμένετε να ακούσετε τι λένε τα 27 διαφορετικά κράτη-μέλη. Μα 27 Υπουργοί Εξωτερικών είναι φυσικό να έχουν και ο καθένας και διαφορετική άποψη ή κάποιες διαφορετικές απόψεις. Εσείς λοιπόν να προσπαθήσετε να πείσετε τους υπουργούς ότι αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα σωστά και αυτά θα πράξει. Συνάδελφο Σούλτς και μετά κυρία Λέζινγκ. Σύντομη, μια σύντομη μάτια και καθυστερημένη για τον συνάδελφο Λάμστορφ. Ήταν μακρύς ο δρόμος και δύσκολος των Γερμανών Πρασίνων από ε, ειρηνιστική θέση σε αυτή τη ε, θέση υποστήριξης ασφαλείας ως εσχάτη λύση παρά αυτή η στάση που είχαν οι φιλελεύθεροι της Γερμανίας της αποχής. Είναι τεράστια η ε, δουλειά που έχετε και είναι και τεράστιες οι προσδοκίες. Πραγματικά κάνετε πολύ καλή δουλειά και ακούω για παρέμβαση, επέμβαση ή όπως είπε ο κύριος ε, Πούτιν για εκστρατεία του ΝΑΤΟ ή για ε, σταυροφορία ε, δεν είναι αυτό που κάνει η Ρωσία σε δύο χώρες σταθμεύουν στρατεύματά της χωρίς εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και στη Γεωργία ε, ο πόλεμος ήταν χωρίς ε, εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην Απχασία και στην Οσετία παραμένουν τα στρατεύματα. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ψήφισμα. Ο κύριος Λαυρόφ σας έχει στείλει μια επιστολή για τη λύση του προβλήματος της υπερνηστερίας. Μπορείτε να μας πείτε τι σας πρότεινε και πώς πρόκειται να ανταποκριθείτε ε, προσεχώς αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόιζα. Και μετά κύριε Κυρία Έστον, η συνάδελφοι, και απευθύνομαι στο Σούλτ και Σύμφωνα με τις εκθέσεις, οι βομβαρδισμοί στη Λιβύη ε, γίνονται πάνω σε καταφύγια, σε ε, αποθήκες όπλων και έχουν καταστραφεί όμως και ε, νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν εσείς λέτε ότι αυτές είναι επεμβάσεις για να επιβληθεί η ζώνη απαγόρευσης πίσω και δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι πρόκειται εδώ για υποστήριξη της μίας πλευράς ε, μιας εμπόλυμης κατάστασης και εδώ θέμα διεθνούς δικαίου και ακόμα και, ακόμα και αν πει κανείς ότι όλα αυτά ε, δικαιολογούνται από το άρθρο 4 του 1973 εγώ ερωτώ ο Αραβικός Σύνδεσμος ε, και η αντιπολίτευση στη Λιβύη δεν είναι εκείνοι που έλεγαν ότι δεν θέλουμε την απαγόρευση αυτή τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων σε προηγούμενες συνεδριάσεις λέγαμε συνεχώς ότι η υποστήριξη του Αραβικού Συνδέσμου είναι καθοριστική σημασία για να υπάρξει επέμβαση. Και κάτι άλλο όσον αφορά τη στρατηγική. Μιλάτε για απελευθέρωση του Λιβικού λαού, μα υπάρχει στρατηγική. Και ποια είναι τα πρότυπα αυτής της στρατηγικής του παρελθόντος, του Ιράκ, τι έγινε τελικά με την απελευθέρωση του Ιρακινού λαού. Αφγανιστάν. Μα τι έγινε με την απελευθέρωση των Αφγανών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, εγώ να ρωτήσω τους σοσιαλδημοκράτες και τους ε, πράσινους ε, Γερμανούς εσείς δεν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσον πράγματι είναι, νομιμοποιείται αυτή η μονομερής παρέμβαση υπέρ της μίας εμπλεκόμενης πλευράς από το διεθνές δίκαιο. Συνάδελφος Μούνης και επόμενος Κόουελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Άστον. Και συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο Υγίστε της ε, αντίδρασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας υποστηρίξω κι εγώ και η Ισπανική Βουλή υποστήριξε την Ισπανική Κυβέρνηση για την εφαρμογή ε, του ψηφίσματος και την εμπλοκή της ε, Ισπανίας με συντριπτική πλειοψηφία 336 υπέρ 3 ψήφοι κατά. Για την Ιεμένη, κυρία Άστον, παρατηρούμε μια κατάσταση που μπορεί να ε, καταλήξει σε μια μετάβαση τύπου Αιγύπτου ή σε πόλεμο τύπου Λιβύης. Οι πρέσβεις της Ιεμένης παρετούνται, εγκαταλείπουν ε, την Ιεμένη, παρετούνται και οι υπουργοί. Ε, πρότεινε ο πρόεδρος το 2012 εκλογές, η αντιπολίτευση απορρίπτει αυτό το μήνυμα αυτό, αυτή την κίνηση τελευταία στιγμή. Οι υπηρεσίες σας έχουν εκτιμήσει ε, την κατάσταση, επεξεργάζονται διάφορα σενάρια, επιζητούν ε, ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για βοήθεια στη μετάβαση σε περίπτωση που θα είναι ειρηνική στην Ιεμένη. Δηλαδή, ε, κάνετε αυτή τη στιγμή προληπτική διπλωματία για να μην επαναληφθεί στην Ιεμένη αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Κόουελ και μετά ο κύριος Χαουίτ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα σε σχέση με την πολιτική μας προς Ανατολάς. Οι γειτονές μας παρακολουθούν πολύ στενά τα όσα κάνουμε για την πολιτική γειτονία. Αναμένουν σαφείς ε, χειρονομίες και μηνύματα. Θέλω να ακούσουν από εμά ότι η πολιτική μας θα έχει περισσότερο στόχο την κοινωνία των πολιτών και ότι θα είναι πιο δραστήρια. Ωστόσο, πέρα από την Ουκρανία, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την ε, Λευκορωσία. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Σικόρσκι πριν από λίγες μέρες είπε ότι μοίρα του κ. Κασιάνκου μπορεί να είναι παρόμοια με αυτή των βορειοαφρικανών σατράπηδων. Αν... Τι πιστεύετε λοιπόν για την Λευκορωσία, οι αντιδράσεις μας είναι ε, τώρα ή θα βρεθούμε ε, με τα όπλα στο χέρι άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χαουίτ και μετά ο κύριος Νεύσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπατεκπρόσωπη. Για τη Λιβύη δεν υπάρχει τίποτα πιο ανθρωπιστικό από το να εξασφαλίσουμε την παροχή νερού στους ε, ανθρώπους που ζουν εκεί. Εσείς μιλήσατε για το δίκτυο επαφών που κάνατε στη Λιβύη, αλλά διαρωτώ με αν είπατε εκπρόσωπος θα μπορούσε να μας δώσει την αξιολόγησή της για το πόσο θα είναι δυνατόν να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διεθνή συνένεση υπέρ της ανθρωπιστικής στρατιωτικής δράσης στη χώρα αυτή και για την Αίγυπτο. Όπως ίσως γνωρίζετε, ήμουν μία από, ένας από τους βουλευτές που ήμουν εκεί για το δημοψήφισμα και στην, ε, μίλησα με αυτούς που ήταν στην πλατεία τα ΓΡΕΚ, τους νέους, και μου είπαν ότι θέλουν περισσότερη δική μας βοήθεια και όχι λιγότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως η προοπτική πρόωρων εκλογών που προβλέπουν, προβλέπεται μέσω του απάντηση στο δημοψήφισμα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να στηρίξουμε τα πολιτικά κόμματα και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο και έτσι επιγόντως να φτάσουμε σε συμφωνία με το Αιγυπτιακό Στρατιωτικό Συμβούλιο σε σχέση με το κατά πόσο θα μπορούμε να στείλουμε μια αναποστολή παρατήρησης των εκλογών για εκλογές μπορεί να γίνουν τόσο γρήγορα όσο, τον, ε, όσο ο Ιούνιος. Ευχαριστώ και ο κύριος Νεύσκη τώρα. Η κυρία Νεύσκη, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Άστον, το ψήφισμα 1973 είναι σαφέστατο μήνυμα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι εσωτερικό ζήτημα μιας χώρας. Η συνένεση στο θέμα αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η Ρωσία, η Κίνα, ακόμα και η Γερμανία, παρακαλώ, δεν έθεσαν βέτο και δεν σταμάτησαν το ψήφισμα αυτό. Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, θα πρέπει να την καλωσορίσουμε. Προφανώς ήταν διαφορετικές οι απόψεις και οι θέσεις. Ωστόσο, εγώ το θεωρώ ως ένα ποιοτικά νέο στάδιο στις διεθνείς σχέσεις. Στη συνέχεια, τον Καντάφη τον υποστηρίζουν χώρες τύπου Λευκορωσίας και Σερβίας. Και αυτό δείχνει ότι δεν είναι μια σύγκρουση εδώ μεταξύ του Ισλάμ και του χριστιανισμού, αλλά είναι ένα ε, πεδίο αντιπαράθεση ε, δημοκρατιών με δικτατορίε. Η στρατηγική μας θα πρέπει να βασίζεται ακριβώς σε αυτό, ιδιαίτερα απέναντι στη Μέση Ανατολή. Επίσης, Μέχρι στιγμής ήταν μάλλον απλουστευτική η προσέγγιση που είχαμε ε, προς τη Μέση Ανατολή, αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ έτσι. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι η Μέση Ανατολή είναι είτε δικτάτορες είτε Ισλαμιστές. Ε, αλλά τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο σχετικά και περισσότερες οι αποχρώσεις και ήταν πολύ σημαντική η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης για τις επαναστάσεις στην περιοχή και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος είναι περισσότερο από ό,τι πετρέλαιο και συμφέροντα. Sorry, thank you. <laughs> Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλη μια, Ρωσία, ε, μια ερώτηση, γνώμη έχω και εγώ, κυρία Εκπρόσωπη, για τη Λευκορωσία. Ε, δύο ψηφίσματα εγκρίναμε φέτος για τη Λευκορωσία. Για να αρχίσουν ε, οι διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων διαβατηρίων. Οι περισσότεροι βουλευτές θεωρούν ότι θα πρέπει να μειωθεί ε, το τέλος αυτό 60 ευρώ για τις χώρες του Σέγγεν. Είναι απαγορευτικό για τους Λευκορώσους. Αν μειωθεί ε, θα βελτιωθεί η κυκλοφορία των ε, πολιτών της Λευκορωσίας και θα γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε θα αρχίσει αυτή η συμφωνία και ποια είναι η στάση της κυβέρνησης της Λευκορωσίας. Ευχαριστώ. Βαρόνι Άστον, έχετε το λόγο για να συνοψίσετε για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω. Πολλές ερωτήσεις έγιναν σε αυτό το γύρο. Όσο μπορώ θα απαντήσω. Κύριε ε, Ρούτσεκ, για τη χάραξη στρατηγικής για τις χώρες του κόλπου, ε, με το Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών, του κόλπου του Περσικού. Έχουμε συνεργαστεί με υπουργού από καιρού καιρών με διάφορους τρόπους. Είναι καλός ο διάλογος που κάνουμε και εκείνοι θα σας πούν πρώτοι ότι θέλουν να τους βλέπουμε ως ξεχωριστά κράτη με ε, το δικό του μέλλον το καθένα και με διαφοροποιημένη αντιμετώπιση, όχι ενιαία. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε. Συμφωνούμε για την Τουρκία επίσης. Η Τουρκία είναι ο πιο σημαντικός εταίρος με τον οποίο συνεργάζομαι με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Κύριε Κούκα, Συμφωνώ απολύτω με αυτά που είπατε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κόσοβο. Όντω δεν είχα απαντήσει. Θα το πω και αύριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σα υπόσχομαι. Και επίση το εμπόριο είναι σημαντικό να αυξηθεί για την ε, Πρίστινα. Και ο Ρόμπερτ Κούπερ ε, το συζητούσε μαζί μου χτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δει το κοσυφοπαίδιο, να καταλάβει ότι αυτός ο διάλογος, ε, αυτές οι επαφές είναι για αυτούς, για το μέλλον τους. Και πραγματικά θέλω να ε, ενισχυθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ε, να έχουν το προσκεκλημένο αυτό. Το ζήτησε η Πρίστινα. Ε, τους εύχομαι κάθε επιτυχία και από τι οφόρο τιμής και στις δύο πλευρές. Κύριε Αρλάκη, το σχέδιο Μάρσαλ. Είπατε ότι χρειάζεται πολλούς πόρους και συμφωνώ. Βεβαίως δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να κατάσχουμε έτσι ε, τα περιουσιακά στοιχεία του κόσμου. Το πάγωμα επιτρέπεται και το κάνουμε. Ε, το θέμα είναι σε ποιον ανήκουν. Αυτό είναι δύσκολο και σημαντικό. Το να έχουμε ε, ευρύ σχέδιο και οικονομικούς πόρους είναι θέμα αναγνώρισης. Ορισμένες χώρες είχαν ε, οικονομικούς πόρους που τους ε, πήραμε. Δεν ξέρω, δεν γίνονται πάντα τόσο εύκολα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε και το εκτιμώ. Ε, στη συνέχεια, για το Ιράν, πότε θα έχουμε τον κατάλογο των προσώπων. Εδώ λέει γρήγορα, <laughs> τον οποίον απαγορεύουμε. Συγγνώμη, δεν ξέρω την ακριβή ημερομηνία από ότι θα καταρτιστεί αυτός ο κατάλογος. Η Ιρανική επιρροή στον Μπαχρέιν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αφενός, δεν θέλω να θεωρηθεί ως λόγος αυτό ε, και δικαιολογία για να μην ε, συνεννοείται με τους διαδηλωτές ε, των Παχρέν. Από την άλλη, οι Αμερικανοί έχουν αρχίσει και ανησυχούν γι' αυτό. Θα πρέπει να ευρεθεί μια ισορροπία, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημαντικός ο διάλογος να προχωρήσει θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό το θέμα σε άλλες ερωτήσεις που έγιναν. Κυρία Νίμπλε, εγώ δεν προσπάθησα καθόλου να ε, διεκπαιρεώσω γρήγορα γρήγορα το θέμα του Μπαχρέιν. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο διάδοχος, ο πρίγκιπας του Μπαχρέιν, προτείνει κάτι ενδιαφέρον για να αρχίσει ο διάλογος, χωρίς προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις, για να ακουστεί όλο το φάσμα των απόψεων. Ε, σιγά σιγά να συμμετέχουν και να υπάρχει ένα είδος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ε, συνταγματικής μοναρχίας, κάτι τέτοιο. Μόνοι τους θα πρέπει να το βρουν. Αλλά έχει ε, ο διάδοχο σχέδιο, αλλά το θέμα είναι να συμμετέχουν όλοι. Γιατί αν υπήρχαν προϋποθέσεις δεν θα συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Να θέλει από μηδενική βάση να ξεκινήσει διάλογος. Αλλά το σημαντικό είναι να προχωρήσει γρήγορα. Μιλήσαμε με τον βασιλικό απεσταλμένο και ε, δηλώσαμε ότι συμφωνούμε. Η ε, βία που έχει εκραγεί είναι πάρα πολύ ανησυχητική ε, και όχι μόνο για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως. Όταν συζήτησα με τον Υπουργό Εξωτερικών του είπα ότι πρέπει να ενημερώσετε τον κόσμο γιατί τι προθέσεις σας και ο Ρόμπερτ Κούπερ το συζήτησε και οι τέσσερις πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν στον Μπαχρέιν από διάφορες χώρες να τους ρωτήσετε, είπαμε, τι θέλουν να γίνει και τους διατηρωτές και να τους συζητήσετε, τι, τι ζητούν, εν πάση περιπτώσει. Και δικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε αυτό το διάλογο. Νομίζω ότι η, η αντιπολίτευση θέλει να αρχίσει το διάλογο και η κυβέρνηση. Το θέμα είναι πώς θα ξεκινήσει αυτό. Υπάρχουν πολλές ιδέες, θα δούμε πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε και ποιο ε, να βοηθήσουμε ε, στη διαδικασία αυτή. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε ε, μια διαφορά στην προσέγγιση μας. Είναι πολύ διαφορετικές οι χώρες, να είναι διαφοροποιημένη προσέγγιση. Άλλο θέλουμε και άλλο θέλει μια χώρα. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθούμε χωρίς να επιβάλλουμε τίποτα. Και αυτό πρόκληση είναι δύσκολο. 27 κράτη-μέλη. Αλλά τι να κάνω εγώ, να έχω την ευρωπαϊκή θέση και να τη λέω στους 27. Έχω συγκεκριμένο έργο, αποστολή και πόρους και για να το κάνω αυτό χρειάζομαι και τα 27 κράτη-μέλη. Και η μεγάλη χαρά, η απόλαυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να συμφωνούν και 27. Η διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή είναι κάτι που αυξάνει το ρόλο μας εκεί, γιατί μιλώ εξ ονόματος 27 κρατών. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα κράτη είναι κυρίαρχα και παίρνουν τις αποφάσεις. Ε, έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ψήφισμα, κανένας δεν το καταψήφισε. Ε, στα συμπεράσματα του Συμβολίου τα υποστήριξαν οι πάντες. Και αυτό δεν είναι ε, απορία άξιων. Γίνεται μεγάλη συζήτηση. Εγώ όμω κάνω τι διερευνητικέ επαφέ, προτείνω, ρωτώ και ζητώ από του σχεδιαστέ να κάνουν το σχεδιασμό και στη συνέχεια ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που αποφασίζει. Εγώ πραγματικά παίρνω πρωτοβουλίες για πολλά πράγματα, αλλά στη τελική ανάλυση, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ε, τα στοιχεία ενεργητικού και τα μέσα που έχουν οι χώρε στη διάθεσή του πρέπει και εκείνες να συμφωνούν. Με ρώτησε ο κύριο Σούλτ για την υπερδνηστερία. Νομίζω ότι είναι ευρεία η συμφωνία για τον απότερο στόχο. Έχω συζητήσει με τους Μολδαβούς υπουργούς πριν από λίγες εβδομάδες και με τους Ρώσους και είναι σαφές ότι θέλουμε να προχωρήσει η υπόθεση εκεί στην υπερδυνστερία. Να κατανοήσει ότι το μέλλον της είναι στη Μολδαβία για κάποια ζητήματα κλειδιά να λυθούν επί τόπου, αλλά μπορεί να συμφωνούμε όλοι για το στόχο. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε ως εκεί. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να συνεννοηθούμε με τη Ρωσία για να προχωρήσει. Κατά την άποψή μου αυτό το πρόβλημα έχει λύση, γιατί ο καθένας ξέρει τι θέλει να κάνει. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο να φτάσουμε ως εκεί. Επίσης είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι έχουμε και πολλά άλλα πράγματα που μας ανησυχούν ε, στο Νότο. Τις επόμενες ε, εβδομάδες θα ε, προσπαθήσω πραγματικά να βοηθήσω. Κυρία Λόιζινγκ, για τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τον Αραβικό Σύνδεσμο και ότι η υποστήριξή του είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, είναι σημαντική, αλλά είναι και πολύ περίπλοκη. Τι κάνουμε εκεί με τη γειτονία. Ό,τι κάνουμε είναι περίπλοκο. Γιατί για κάθε χώρα τα προβλήματα είναι περίπλοκα και θα πρέπει και να τα αναγνωρίσουμε και να τα σεβαστούμε. Δεν είναι απλώς ένα θέμα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, στην Αίγυπτο, την Τινησία, στον Μπαχρέιν, αλλά να αναγνωρίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε για το λαό με τον πιο αποτελεσματικό κόπο, τρόπο. Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα και είναι περίπλοκο. Όταν γυρίσαμε από τις διακοπές των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά, κανένας δεν είχε προβλέψει την κατάσταση που είμαστε τώρα. Πριν από 6-8 εβδομάδες δεν είχαμε ιδέα. Θα μπορούσα να σας πω ποιες χώρες με ανησυχούσαν τότε. Θα ήταν το Σουδάν, οι ακτέρα φανταστούν ακόμα με προβληματίζουν, αλλά δεν ήξερα ότι θα βρισκόμασταν τέτοιες ώρες εδώ να λέμε αυτά που λέμε. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τους λαούς αυτών των χωρών και να συνεργαστούμε. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός ο αραβικός σύνδεσμος και γι' αυτό βρισκόμαστε σε διάλογο μόνιμο και με τον Άμρα Μούσα. Μιλήσαμε και σήμερα και το Σαββατοκύριακο και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σε επαφή. Και έχω τεράστιο σεβασμό για το έργο του αραβικού συνδέσμου. Δεν νομίζω ότι διαφέρουν για την Ιεμένη. Όπως τη βλέπουμε τώρα, ανταποκρίνεται στα όσα φοβόμουν, στους χειρότερους φόβους μου. Τους τελευταίους μήνες είδαμε και τον πρόεδρο Σαλέχ και υπουργού και προσπαθήσαμε να τους πούμε να έρθουν σε επαφή σε εθνικό διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό έχω καταλάβει ότι θέλει αντιπολίτευση. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε τώρα να βεβαιωθούμε ότι θα εξακολουθήσουμε να τους πιέζουμε. Τώρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Ο πρόεδρος είπε, ε, ε, πρότεινε κάτι να αποσυρθεί, αλλά το, το απέρριψε η αντιπολίτευση, αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα. Ε, θα πρέπει να τα παρακολουθούμε πολύ στενά, είναι πολύ ανησυχητικά και πραγματικά ε, η πραγματικότητα έχει επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους μου. Η πολιτική γειτονία θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένη, ναι, για να μπορεί να αντιδρά πιο γρήγορα, πιο διαφοροποιημένα, πιο ευέλικτα, να αναγνωρίζει τι πρέπει να γίνει σε κάθε χώρα και να μπορεί να κινητοποιεί και τους πόρους το συντομότερο επιτόπου. Θα πρέπει να είμαστε και πιο γρήγοροι και καλύτεροι και πιο έξυπνοι στα όσα κάνουμε. Για τη Λευκορωσία. Εχθές το συζητήσαμε για να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε και τα μέτρα αυτά. Συνάντησα τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσίας ε, καθώς έβγαιναν από τη φυλακή ή με εκπροσώπους τους της οικογένειάς τους, πραγματικά συμφωνούν όλοι ότι είναι φρικτή η κατάσταση και κάναμε διαβήματα και στον κύριο Μαρτίνοφ του ξεκαθάρισα τι περιμένουμε από τη χώρα να κάνει, αλλά ανησυχώ. Δεν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Για το συνδυασμό, περιοριστικά μέτρα, αλλά και διατήρηση διαλόγου με το λαό της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χάουιτ με ρώτησε για τη διεθνή συνένεση. Βεβαίως είναι σημαντική, αλλά είναι και δεδομένη. Συνεργάζονται όλοι από διάφορα πρίσματα, στενά όμως, με διάφορους τρόπους. Οι νέοι θέλουν περισσότερη Ευρώπη, συμφωνώ. Ε, και, και οι αραβικοί λαοί θέλουν μεγαλύτερη υποστήριξη. Ε, είναι πρόκληση οι εκλογές τώρα και οι νέοι της Αιγύπτου ανησυχούν και ε, θεωρούν ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά θέλουν, ε, θέλουμε να μας καλέσουν κιόλας ε, για την υποστήριξη εκλογές. Προσπαθήσαμε να το παρακολουθήσουμε ε, και το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Η κυρία Νεύσκη, για την απλουστευμένη, απλουστευτική μάλλον προσέγγιση που είχαμε λέτε στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω με τον τρόπο που τα παρουσιάζετε τα πράγματα εγώ. Ε, βλέπουμε ε, το θέμα αυτό σαν παροδία ε, ότι διάφορες παραδόσεις έχουν διαφορετικές αξίες. Δεν είναι ευρωπαϊκές αξίες αυτές και οι αρχές είναι παγκόσμιες. Να μην είμαστε υπερβολικά απλουστευτικοί στον τρόπο που το κάνουμε όμως. Για τη Λευκορωσία, κύριε Παλέσχης, ορίσαμε τη διαπραγματευτική εντολή για τη διευκόλυνση θεώρηση διαβατηρίων στις 28 Φεβρουαρίου και αποσκοπούμε στην έναρξη των συζητήσεων. Ξέρετε ότι δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, μακρηγόρησα πάρα πολύ. Δεν το έκανα και εμένα. Ε, και ε, περίμενα να με ρωτήσει κάποιος γιατί δεν ασχολούμαι με λιγότερα. Δεν το έκανε κανείς. Δηλαδή, φανταστείτε να σας έλεγα ότι όχι, δεν θα ασχοληθώ με το τώρα, θα κάνω λιγότερα. Είναι πραγματικά σαν να πετάς ένα αεροπλάνο όταν σου ε, κολλάνε τα φτερά εκείνη την ώρα και κάποιος ταυτόχρονα προσπαθεί να κόψει την ουρά του αεροσκάφους. Είναι δύσκολη προσπάθεια, αλλά εμείς θα εξακολουθήσουμε να προχωρούμε προς την κατεύθυνση αυτή και είναι μεγάλη τιμή για μένα να το κάνω αυτό εξ ονόματός σας και των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε και άλλη μια φορά ε, κύριε Πατεκπρόσωπο και ελπίζουμε να σα δούμε πιο σύντομα με λιγότερα προβλήματα. Συνάδελφοι, μην απομακρύνεστε γιατί θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κύριε Τάνοκ. Colleghi, Συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. για την πρόταση ψηφίσματο για την έκθεση που αφορά την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ισλανδία του 2010. Η ο κ. Κρίστιαν Πρέντα. παρακαλώ λοιπόν να τοποθετήσετε στη σχισμή την κάρτα σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ε, συμφωνείτε να προχωρήσουμε. Παράγραφος 3, τροπολογία 1. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Σας παρακαλώ να ψηφίσουμε για το πρώτο τμήμα.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 Προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 3 υπέρ κατά. Σας παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια σας. Ποιοι είναι υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 13, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Στο δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική. Περθών 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 γιατί η 16 έχει καταπέσει. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Σας ζητώ να ψηφίσετε. Sì. Chiudiamo Τέλος ψηφοφορίας, αν και κάποιος που δεν θέλει να ψηφίσει. Υπέρα. με μεγάλη πλειοψηφία, εγκρίνεται. Ευχαριστώ.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 Συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον με την εξέταση της κατάστασης στο βασίλειο του Μπαχρέιν. Υποδεχόμαστε τον κύριο Μιγκαρέλη καθώς και τον κύριο Κούπερ που πήγαν στο Μπαχρέιν ως εκπρόσωποι της ύπατας εκπροσώπου και φυσικά έχουμε μαζί στο Πραδείο του κυρία Αγγέλικα Νίμπλερ που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για το Περσικό Κόλπο. Κύριε Μιγκαρελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πάντα χαίρομαι όταν με καλείτε για να ε, σας παρουσιάσουμε τις αναλύσεις μας και ε, τις θέσεις μας στους βουλευτές. Το Παχρέιν γνωρίζετε τα γεγονότα, δεν έχουμε επιτόπου αντιπροσωπεία και ε, επαφή έμεθα στα όσα μας λέει ο πρέσβης μας που είναι στο Ριάτ, στη Σαουδική Αραβία και διαπιστευμένος και στα υπόλοιπα κράτη του Περσικού Κόρπου και ακούμε και από τις πρεσβείες των κρατών μελών όσα μας αναφέρουν. Εδώ και κάποιες εβδομάδες έχει ξεσπάσει μια σύγκρουση μεταξύ της ε, πλειονότητας του πληθυσμού που εκφράζει πολιτική, κοινωνική και οικονομική απογοήτευση και, τους και των ηγετών της χώρας αυτής. Ε, φαίνεται και τονίζω ότι φαίνεται ότι ε, οφείλεται αυτό, αυτή η δυσφορία και η ε, απογοήτευση στην αρχή ήταν μόνο οικονομική, πολιτική και κοινωνική. Δηλαδή η πλειονότητα του πληθυσμού θεωρούσε ότι το καθεστώς δεν ε, διένει με τον πλούτο της χώρας ε, τον πληθυσμό αυτό και από πολιτικής απόψεως οι αποφάσεις λαμβάνονται από μία μειοψηφία, μειονότητα και δεν γινόταν ε, σεβαστή η πλειονότητα του πληθυσμού και ε, πολύ γρήγορα ε, αυτό πήρε θρησκευτικό χαρακτήρα. Γνωρίζετε ότι 70% είναι οι Σιήτες στη χώρα και 30% Σουνίτες. Και εκεί περιπλέκονται βεβαίως τα πράγματα. Στην αρχή και αυτό που συστήσαμε αμέσως στις αρχές ήταν να προσπαθήσουν να προβούν σε γνήσιο ειλικρινή διάλογο με τους ε, διαδηλωτές για να προσπαθήσουν να ε, ανταποκριθούν στις αρχικές τους ε, διεκδικήσεις οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα. Να συμμετέχει στον πολιτικό βίο της χώρας, δηλαδή του βασιλείου, μεγαλύτερος ε, αριθμός ε, πολιτών. Ποτέ όμως δεν άρχισε αυτός ο διάλογος και σιγά σιγά φαίνεται η σύγκρουση αυτή η οποία ε, φρονώ ότι στην αρχή ήταν κοινωνικού χαρακτήρα, πήρε ένα όλο και περισσότερο θρησκευτικό χαρακτήρα. Και εδώ βεβαίως τα πράγματα περιπλέκονται και γίνονται και πιο ευαίσθητα γιατί ε, έχουμε μεγαλύτερες περιφερειακές επιπτώσεις. Είναι σαφές ότι μια πλειονότητα Σιητών που θεωρεί ότι καταπιέζεται στο Μπαχρέιν θα έχει σημαντικές ε, συνέπειες και στο Ιράκ όπου γνωρίζεται η πλειονότητα η Σιητική σήμερα προσπαθεί να ε, ανακτήσει μια ισορροπία στη διαχείριση της εξουσίας με τους Σουνίτες, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό. Επίσης έχει επιπτώσεις και στο Λίβανο, όπου είχε πολλά ε, εκδήλωσε την αλληλεγγύη και τη συμπάθειά του προς τη σιητική πλειονότητα του Μπαχρέιν και βεβαίως υπάρχει και μειονότητα σιητική στην Ανατολική Σαουδική Αραβία στην περιοχή που είναι τα κοιτάσματα των υδρογών ανθράκων. Είναι λοιπόν η κρίση εσωτερική στο Μπαχρέιν ε, ταυτόχρονα που επιδεινώθηκε ακριβώς επειδή δεν δείχνουν οι αρχές της χώρας καμία βούληση, καμία πρόθεση να αρχίσουν ένα γνήσιο εθνικό διάλογο και υπάρχει και η περιφερειακή διάσταση γιατί αν αυτά ε, οδηγηθούν σε θρησκευτική σύγκριση, υπάρχουν χώρες της Μέσης Ανατολής που ε, κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες. Απέναντι σε αυτά είπα τι εκπρόσωπος τηλεφώνησε ε, στον Υπουργό Εξωτερικών για να τους ζητήσει να ε, δείξουν συγκράτηση οι δυνάμεις τάξεως, να μην χρησιμοποιήσουν τη βία, για να προτείνει να αρχίσει ένας εθνικός διάλογος. Επίσης δήλωσε η κυρία Στον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να διευκολύνει την κατάσταση αν μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Έστειλε και το Ρόμπερτ Κούπερ στη χώρα πριν από λίγες μέρες η κυρία Στον και ακολούθησε χθεσινή δήλωση Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που με δύο λόγια καταγγέλει τη βία των τελευταίων ημερών, ε, απευθύνει έκκληση και στις δύο πλευρές προς συγκράτηση αλλά κυρίως προς τις εθνικές ε, αρχές, ε, ζητεί την έναρξη εθνικού διαλόγου και βεβαίως κατά κάποιο τρόπο προσφέρει τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά μπορεί κανείς να πει αυτή τη στιγμή για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Στις Βρυξέλλες ε, εδώ και λίγες εβδομάδες ε, έχει έρθει και ένας εκπρόσωπος του βασιλιά, του Μπαχρέν. Τον συναντούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει πραγματικά στη χώρα. Αυτά ήθελα να σας πω. Στις 20 Απριλίου συνεδριάζει ετήσια διυπουργική συνέλευση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα έχουμε την ευκαιρία να ε, περάσουμε κάποια μηνύματα. Τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, τα μέσα δράσης και η μοχλή που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένη και πίεσης. Και όπως γνωρίζετε, τα ουδαραβικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί στο Μπαχρέιν και κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο ευαίσθητη. Αυτά με δύο λόγια νομίζω συνοψίζουν τη σημερινή κατάσταση στον Παχρέιν. Στο κύριε Κούπερ θέλετε να προσθέσετε κάτι Α, αργότερα. Εντάξει. Νίπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μόνο τρεις ε, παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή που ε, θεωρεί το θέμα του Μπαχρά ένα σημαντικό θέμα, το βάζει στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ που ήρθατε εσείς ε, και που οι εμπειρογνώμονες επίσης θα μας δώσουν και τις απαραίτητες πληροφορίες. Δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να διεξάγει διάλογο και από ό,τι άκουσα όμως ο διάλογος αυτός τελικά δεν έλαβε χώρα. Ε, ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε ο διάλογος και να μας πείτε και μία προσωπική σας ε, γνώμη. Υπάρχει περίπτωση να επανέλθει, να εντατικοποιηθεί ο διάλογος, γιατί νομίζω ότι μόνο αυτή τη δυνατότητα έχουμε ε, έτσι ώστε να φέρουμε κάποια κίνηση σε θέματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Και δεύτερο ερώτημα, δεν είπατε ότι η κυβέρνηση του Μπαχρέιν ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία στρατιωτική ε, συνδρομή. Ίσως ε, να ήτιστε εκεί στην περιοχή όταν έχει κάποιος πρόβλημα να ζητάει τη στρατιωτική ε, σύνδρομη μιας γειτονικής χώρας. Και μέσα από το ε, διαδίκτυο έχω και εγώ πολλές ειδήσει από γνωστούς ότι στην περιοχή και ασκείται βία, εκτεταμένη βία. Πήρα λοιπόν πολλά email που μου επισημαίνουν ότι ο κύριος Ναμπίλ Ράγιαπ αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρόεδρος ε, του Κέντρου του Μπαχρέν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνελήφθη. Μήπω μπορείτε εσεί να πείτε κάτι από αυτού. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι μεμονωμένη περίπτωση, γιατί και διαδηλωτέ ε, που διαδήλωναν ε, ειρηνικά και αυτοί συνελήφθησαν. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε από εσά από πρώτο χέρι ποια είναι η αξιολογησή σα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι. Και τελευταία ερώτηση. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να εμβαθύνετε στο ποιες ε, επιπτώσεις θα έχει η κατάσταση στο Μπαχρέιν σε όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Και επειδή εσείς έρχεστε από την περιοχή, μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Ah, Θέλω να σας θέσω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζήτησα πριν από την είπατε εκπρόσωπη να μην ε, έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά, διαφορετικά μέτρα και σταθμά και να καταδικάσει το σπυραβαλισμούς ε, κατά των διαδηλωτών ε, γιατί η στάση της κυβέρνησης ήταν ε, πολύ έντονη σε σχέση με τους διαδηλωτές ανεξάρτητα που είναι, που είναι σύμμαχός μας τον Παχρέιν και είναι και η έδρα του έκτου στόλου το Αμερικανικό εκτοστόλου. Φαίνεται όμως να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του, και του Βασιλιά. Ο Πρωθυπουργό φαίνεται να, να περνάει το δικό του περισσότερο και σίγουρα δεν έχει κάνει και πολλά ο για να ανέλθει η πλειοψηφία των ε, Σουνιτών. Ε, και μάλιστα τελευταία διάβασα ότι είναι δύσκολο να βρει κανείς δουλειά εκεί Ακόμα αν δεν είναι από το Βαχρέν. αυτό νομίζω από μόνο του λέει πολλά. Επίσης ανησυχώ για την ε, ιρανική ανάμεξη συμπεριλαμβανομένων απειλών για αναβίωση του, του, των εδαφικών διεκδικήσεων. Είναι κάτι το οποίο ε, ίσως ο Ρόμπερτ Κούπερ θα μπορούσε να απαντήσει, γιατί νόμιζα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όταν αποαπικιοποίησε το Ιράκ είχε μια συμφωνία που είχε γίνει αποδεκτή. Ε, αν και και έπρεπε η Τεχεράνη με βάση αυτή τη συμφωνία να αναγνωρίσει για πάντα την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Μπαχρέιν. Κύριο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μάθαμε ότι ο υπατοσαρμοστής του ΕΣ ΕΕ στη Γενέβη είπε ότι έχουν εξαφανιστεί τις τις εβδομάδες στο Παχρέν 50 με 100 πολίτες μετά από την καταστολή ε, της ε, διαδήλωσης της Τετάρτης. Ε, στο νοσοκομείο της Αλμανίγιας συνέλαβαν γιατρούς, νοσηλευτές. Ε, είναι στη μανά μας την πρωτεύουσα αυτό το νοσοκομείο, το, το οποίο είναι πολύ περίπλοκος προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιδεινώνεται από την εισβολή, γιατί εισβολή τη θεωρώ εγώ της Σαουδικής Αραβίας, Αυτόν αυτής της απολυταρχικής ε, βασιλείας και της φεοδαρχικής ε, μορφής ε, του κράτους της Σαουδικής Αραβίας. Εγώ δεν επιθυμώ στρατιωτική επέμβαση δυτική ούτε στη Σαουδική Αραβία ούτε στον Μπαχρέιν. Γι' αυτό η προηγούμενη τοποθέτησή μου ε, στην κυρία Άστον έλεγε ότι είμαστε υποκριτικοί και άνηση ε, στις συγκρούσεις στον κόσμο. Η Αλ-Σαούντι δυναστεία που βασιλεύει η Σαουδική Αραβία τι έχει. Δεν έχει ούτε κόμματα, ε, ούτε εκλογές, σωματική σοφρονισμοί, κόβουν χέρια, κόβουν πόδια. Η Επιτροπή Βασανιστήριων του ΟΗΕ ε, τα καταδίκασε και οι Σαουδάραβες που έχουν αυτή τη στιγμή πάνω από χίλιους στρατιώτες στο Μπαχρέιν για να βοηθήσουν στην καταστολή, τι απαντούν ότι αυτές οι πρακτικές είναι τμήμα λέει της ε, Ισλαμικής παράδοσης εδώ και 1400 και πλέον έτη για να μην μιλήσω και για την πολιτική της θρησκευτικής αστυνομίας ηθών που επιτηρεί τις γυναίκες να είναι σωστά αντιμένες και όχι μόνες τους ε, στα ε, δημόσια μέσα μεταφοράς να είναι κάποιος άντρας πάντα από την οικογένειά τους είτε ο σύζυγος είτε αδελφός και εφαρμόζουν και τη σαρία. Αυτό είναι λοιπόν το τοπίο κυρίες και κύριοι και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τώρα να επέμβει. Τώρα. Το είπα και πριν την κρίση της Λιβύης, πριν γίνει αυτή η καταστολή και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά τι συμβαίνει. Το πρόβλημα ξέρετε είναι το πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχουμε τώρα με την κρίση τη Λιβύη. Και προφανώ ε, δεν μπορούμε τώρα να στεναχωρήσουμε και μια περιοχή που είναι σημαντικότατη για το πετρέλαιο. Εγώ όμω δεν κάνω διακρίσει και η πολιτική μου ομάδα ούτε βάζει πρώτα τα οικονομικά συμφέροντα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν το κάναμε ούτε με τη Λιβύη ούτε τώρα. Ούτε θα ζητήσουμε όμω στρατιωτική επέμβαση, διότι πρέπει να λυθεί το θέμα δια της διπλωματικής οδού και δια της απέτηση εδώ και τώρα ισχυρή απέτηση να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Μπαχρέν και στη Σαουδική Αραβία. Γνωρίζω ότι είναι φωνή όντω εν τη ερήμο, στο όρο Σινά συγκεκριμένα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δρά έτσι. Δεν δρά έτσι δυστυχώ. Ούτε το έπραξε με τον Μπεναλή αυτό, ούτε με τον Μουμπάρακ, ούτε πρόκειται να το κάνει τώρα. Ούτε το κάνει στον Μπαχρέιν, ούτε στη Σαουδική Αραβία. Και προτιμούμε να έχουμε καλή σχέση με ένα φεοδαρχικό σύστημα που έχει σωματικές τιμωρίες και σοφρονισμούς. Μην τους ενοχλήσουμε και μας κόψουν και το πετρέλαιο και το αργό και τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να ε, μετακινούμαστε ή να έχουμε πετρέλαιο για τις ε, Βιομηχανίε μας. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να έχουμε μια δραστήρια στάση ενεργητική και να δώσουμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο για τα όσα συμβαίνουν στο Μπαχρέν και τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα, εγώ λέω, και τα νέα που μαθαίνουμε, ειδήσει τελευταίε σημερινέ από τη Γενέβη, από την Υπατερμοστία, θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να απαντήσουμε γρήγορα. Αν δεν έχουμε γραφεία, να στείλουμε αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου, του πιο υψηλού επίπεδου που έχουμε στην περιοχή ακριβώς. Να παρατηρήσει εκ του σύνεγγυς τι συμβαίνει και να έχουμε ε, από πρώτο χέρι πληροφορίες που να μπορούμε να τις διασταυρώσουμε, να τις εξακριβώσουμε για να μην πέσουμε τώρα σε μια κλιμάκωση ε, της καταστολής που θα μας οδηγήσει σε πολύ χειρότερες ε, καταστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ σύντομα να ρωτήσω κάτι για τον Μπαχρέιν. Ο συνάδελφος κύριος ε, Λάμστορφ ε, αναφέρθηκε στην κριτική του μηνύματος κυρίας Άστον ε, ζητούσε και τις δύο, ε, τις δύο πλευρές να ε, επιδείξουν συγκράτηση και να σταματήσουν τη βία. Πολύ περίεργα είναι αυτά. Από τη μια έχουμε πολύ καλά οπλισμένες δυνάμεις με ελεύθερους σκοπευτές, με στρατιώτες, αοδάραβες και από την άλλη είναι οι διαδηλωτές. Πού είναι οι ίσες αποστάσεις εδώ. Μου φαίνεται κάπως, πώς να το πω, ανάρμοστο. Και θα ήθελα να μας εξηγήσετε Πώς φτάσατε σε αυτή την εκτίμηση. Επίσης, άλλη μια ερώτηση για τη Σαουδική Αραβία. Τι κάνετε ε, για την επέμβαση αυτή. Τι κάνει το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, πώς το αξιολογεί, ποιες συνέπειες θα έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Chris Kreisel Dörfler, κύριε Μιγκαρέλη, Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για αυτά που είπατε. Ε, είχαμε μια συζήτηση με την κυρία Άστον και εσείς έρχεστε από εκεί, από την περιοχή που επισκεφτήκατε. Πιστεύετε ότι μπορούν να υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ε, δεν ξέρω, είναι βέβαια δύσκολο να πείτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα να το μεταγίνει στη Λιβύη, αλλά εγώ ερωτώ, ε, μήπως ε, η εξέγερση στο, στη Λιβύη προκαλέσει ντόμινο στο Μπαχρέιν που δεν θα ε, ικανοποιηθούν με ελάχιστα ψυχία αλλά θα θέλουν και δικαίως να αποκτήσουν περισσότερα. Εσείς ε, θεωρείτε ότι χρησιμοποιούμε και εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ε, γιατί το γεγονός ε, ότι υπάρχει η Σαουδική Αραβία και εκεί πράγματι υπάρχει μεγάλη συνεργασία με τις ΗΠΑ και ο λιμενισμός του έκτου στόλου. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός, μόνο που πρέπει να προσέξουμε. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας είπα, εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι άλλα πράγματα εφαρμόζουμε στη μία χώρα και άλλα στην άλλη. Τι έχετε να μας πείτε από αυτού. Κυρία Γκόμες. την, Κυριακή, συγγνώμη, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την προεδρία του κ. Μπουζέκ όταν ε, τελειώσαμε ε, τη συνάντηση με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Δεν μπορέσαμε να βγούμε από την κύρια είσοδο, αλλά από μία πλαϊνή, γιατί υπήρχαν νέοι ε, που διαδήλωναν και ζητούσαν δράση κυρίως για την Ιεμένη. Ό,τι λοιπόν και αν κάνουμε η διεθνής κοινότητα και οι κύριε Ευρωπαϊκή Ένωση, μα ό,τι και αν δεν κάνουμε, παρατηρείται, το παρατηρούν, το διαβάζουν, το διαβάζουν οι άνθρωποι τους οποίους υποτίθεται ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε ε, τους ανθρώπους ε, που επιθυμούν τη δημοκρατία στην ε, Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Θα ήθελα να ρωτήσω τους κυρίους Μιγκαρέλη και Κούπερ κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι με τη δήλωση για τον Μπαχρέιν. Μα ποιος την έκανε αυτή τη δήλωση. Πιστεύετε ότι η δήλωση αυτή δείχνει κάποια συνέπεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως ε, κι εσείς ε, πιστεύετε ότι πρόκειται για ένα παραπροϊόν, ε, ένα αποτέλεσμα της διαφωνίας που επικρατεί ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Άλλη μια ερώτηση του κυρίου Φόξ και μετά απαντήσει ο κύριος Μιγκαρέλη. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη του πάνελ για την άποψή σας. Ο συνάδελφος εδώ εκ δεξιών καθήμενος ε, χαρακτήρισε ε, εισβολή της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι υπερβολικό σε μεγάλο βαθμό. Εγώ νομίζω ότι τους κάλεσε η κυβέρνηση του Μπαχρέιν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Και το δεύτερο, σε ποιο βαθμό το Ιράν συμμετέχει στην κατάσταση αυτή. Ε, ε, υποκίνησε τους αντιφρονούντες. Καταλαβαίνω ότι είναι θεμητά τα αιτήματά τους, αλλά εσείς νομίζετε ότι αυτό το υποκίνησε μια ξένη δύναμη. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε με αυτή την πρώτη σειρά ερωτήσεων, να θέσω κι εγώ μία ερώτηση. Είδαμε τα γεγονότα στην Τινησία, στην Αίγυπτο και στη Λιβύη την τηλεόραση Αλτζαζίρα η οποία έδινε ανταποκρίσεις για τις επαναστάσεις και αμφισβητώντας πολύ έντονα τις, ε, τα καθεστώτα. Θα ήθελα να ξέρω πώς ανέφερε τα γεγονότα στο Μπαχρέιν η ίδια τηλεόραση Αλτζαζίρα, στις γειτονικές χώρες όπως το Κατάρα που εδράζεται η Αλτζαζίρα ήταν υπέρ των επαναστατών, των διαδηλωτών ή ήταν πιο ισορροπή η στάση τους. Και πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι στις ε, δυνάμεις που μπήκαν στο Μπαχρέν κατά των διαδηλωτών είναι οι Σαουδάραβες και ε, οι ε, πολίτες των Εμμυράτων, αλλά όχι από το Κατάρ που αντιθέτω είναι στι ε, συμμετέχουσε αποστολέ κατά του Καντάφη στη Λιβύη. Να πω δύο λόγια καταρχήν. Εγώ πιστεύω πως είναι σωστό που το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει αυτό το θέμα και που το εξετάζει σοβαρά. Όλοι θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Γιατί κατά τη διάρκεια της σύντομης περίοδου που επισκέφθηκα τον Μπαχρέιν εξ ονόματος της ΥΠΑ ΕΕ, της αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η πολύ γρήγορη πόλωση της κοινωνίας και έλλειψη διαλόγου βεβαίως. Και ακούγοντας τις δύο πλευρές, γιατί άκουγα, δεν ε, θέλησα εγώ να κάνω τον έξυπνο ή να συμμετέχω στη ζήτηση, φαινόταν να γίνεται διάλογος ε, κοφών. Εγώ εξέφρασα την επιθυμία μας να επανέλθει το Μπαχρέν στην κανονική του κατάσταση, δηλαδή να γίνει και πάλι ένα ειρηνικό ευχάριστο μέρος. Το τελευταίο καιρό υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα είναι μάλλον έκτακτα. Και δεν είμαι βεβαίω ότι χρειάστηκε παλιότερα η αστυνομία του Μπαχρέιν να ασχοληθεί με θέματα τήρησης της τάξη. Δεν είναι εύκολο ε, όταν έχει κανεί αντιμετωπίσει μεγάλες κλίμακε διαδηλώσει ότι μπορεί να ασχηθεί η βία είναι δύσκολο για την αστυνομία, δεν είναι κάτι που τα καταφέρνουμε κι εμεί πολύ καλύτερα ακόμα και στι καλύτερε δυτικέ χώρε. συμβαίνουν ατυχήματα και μάλιστα η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η αστυνομία μία από αυτές τις διαδηλώσεις. εν πάση περιπτώσει είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η μόνη βία μέχρι στιγμής ήταν από πλευράς των, της αστυνομίας και των αρχών. Υπήρξε και ασκήθηκε βία και από κάποιους από τους διαδηλωτές και υπήρξαν και θάνατοι τουλάχιστον δύο αστυνομικών. Επίσης, υπήρξε βία από διάφορες ένοπλες ομάδες που ήταν εκτός ελέγχου, οποιοδήποτε ελέγχου. Και από τις δύο πλευρές Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κρίνει κανείς ή να κρατηθούν ισορροπίες. Και σε αυτό το πνεύμα το Σύμβολο εχθές ζήτησε από όλε τι πλευρέ να σταματήσουν τη βία. Γιατί φαίνεται... Φαίνεται να υπάρχουν διάφοροι ανεξάρτητοι ε, ανεξάρτητες ομάδες και ανεξέλεγκτες ομάδες οι οποίες ε, συμπεριφέρονται πολύ βία, πολύ δυσάρεστα πράγματα παρόμοια με αυτά που συνέβαιναν παλιότερα στα Βαλκάνια. Τελευταίος ομιλητή ο κύριο Φόξ, είχε δίκιο. Νομίζω εκείνο είπε ότι η τα στρατεύματα της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων ε, ε, ήταν παρόντα μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης ε, του Βαχρέν και νομίζω και κάποιοι κουβειτιανοί. Δεν ήταν ορατοί, δεν συμμετείχαν στον έλεγχο των διαδηλώσεων, των αναταραχών. Από ό,τι κατάλαβα ε, ρόλος τους ήταν να φυλάσσουν κάποιες ε, κύριες εγκαταστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αόρατοι. Ήταν εκεί αλλά χωρίς να παρεμβαίνουν. Οπότε είναι λάθος να υποδίδουμε περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που έχουν πραγματικά αυτές οι δυνάμεις. Για το θέμα του Ιράν, ως ήθιστε με τέτοια θέματα, είναι δύσκολο να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η θέση του Ιράν. Θα ήταν ε, έκπληξη για μένα αν οι Ιρανοί δεν είχαν εντοπίσει ότι υπήρχε εκεί μια σπουδαία ευκαιρία για αυτούς και δεν το είχαν εκμεταλλευτεί. Από την άλλη πλευρά, επίσης δεν ξέρω αν θα έχουν και τόσο υποστηρικτέ στο Μπαχρέιν, ούτω ή άλλω Ιρανοί, γιατί πολύ αμφιβάλλω αν θα επιθυμούσαν καθεστώ παρόμοιο με αυτό το Ιράν. Εκεί. Ίσως αυτό το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό είναι ότι υπήρχε σαφής επιθυμία ανάμεσα στον κόσμο με τον οποίο εγώ συνομίλησα, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Υπήρχε σαφής επιθυμία να ε, ξανακάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου. οι προτάσεις του διαδόχου νομίζω είναι ακόμα επιτάπητος, συζήτηση. αλλά σταμάτησαν να είναι το κύριο σημείο της ημερήσιας διάταξη τη στιγμή που η βία στους δρόμους ε, γενικεύθηκε. Τώρα έχει γίνει μια, ένα διάλειμμα, από ό,τι κατάλαβα η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ήρεμη και νομίζω πως αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να ξεκινήσει ο διάλογος. Ε, η κατάσταση από την άποψη της διαχείρισης του Μπαχρέν που είναι ένα μικρό νησί είχε γίνει σχεδόν ε, αβάσταχτη γιατί συνάδελφος ε, χρειάστηκε τρεις ώρες να φτάσει από το αεροδρόμιο στην πόλη. Αν γνωρίζει κανείς τον Παχρέν, καταλαβαίνει τι σημαίνει κάτι τέτοιο όσον αφορά τα μπλόκα στον δρόμο. Δεν ήταν κίνηση, ήταν μπλόκα. Ένα σωρό κόσμο, όποιο του κατέβαινε, έκανε ένα μπλόκο στο δρόμο. Δεν ήταν ε, ούτε πάντα κυβερνητική, ούτε πάντα η αντιπολίτευση. Οι αρχέ είχαν δίκιο λοιπόν να θέλουν να επιβάλλουν και πάλι την ηρεμία και την τάξη. Αλλά αυτό φυσικά είναι σωστό μόνο αν ανακολουθηθεί από διάλογο και αν οι προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο διάδοχος είναι εξαιρετικές και αποτελούν πολύ καλή βάση ώστε οι δύο πλευρές να κάτσουν και να συζητήσουν. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο για την ώρα και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Εγώ να σε πληρώσω με δύο λόγια για το ρόλο του Ιράν, κύριε Φόξ, δεν είναι απίθανο το Ιράν να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο την κατάσταση, αλλά νομίζω πως θα ήταν μέγα σφάλμα να αποδώσουμε το αίτιο των αναταραχών σε αυτή τη χώρα σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Όχι, δεν ε, λύνονται έτσι τα εγχώρια προβλήματα και έπειτα στη συνέχεια να υπάρξει απόπειρα εκμετάλλευση ε, είναι προφανές. Τώρα για τις συνέπειες για την ε, πολιτική στις υπόλοιπες χώρες. Αν θα προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις, ναι, αναμφίβολα. Δεν υπάρχει ούτε μια αραβική χώρα που να μην έχει επηρεαστεί με κάποιον τρόπο από τα όσα συνέβησαν στην Τινησία, στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Εγώ λοιπόν δεν έχω παρά ελάχιστες αμφιβολίες ότι με ιδιαίτερε βέβαια διαδικασίες σε κάθε μια από τις χώρες οι αθηνικές αρχές ακόμα και αν δεν διαπνέονται σε ορισμένε χώρες από ε, δημοκρατικούς προβληματισμούς θα πρέπει πάντως θα υποχρεωθούν να προβούν σε εξυγχρονισμό της κοινωνίας και να προβούν σε μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένας, ένας άνεμος μεταρρύθμισης που ε, σαρώνει όλες τις χώρες αυτές. Και βέβαια αυτό όχι μόνο στην περιοχή. Εμεί βέβαια τι αρχέ μα περισσότερο με ανθρώπου που είναι αδύναμοι, που δεν έχουν πόρου, παρά με ισχυρού που έχουν πόρου. Και αυτό είναι ισχύει όχι μόνο για αυτή την περιοχή του κόσμου, αλλά για όλε τι περιοχέ του κόσμου. Κύριε Μπραντνερ, τώρα αν θα πρέπει να βάλουμε Επίση, όλου τους διαδηλωτέ και τις δυνάμεις τη τάξη, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι στα ανακοινοθέντα μα θα πρέπει να ζητάμε από τους ε, διαδηλωτέ να αποφύγουν την προσοχή στη βία και έχετε δει και όταν υπάρχουν δεκάδε νεκροί δεν μπορούμε να τους βάλουμε στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο με τις δυνάμεις καταστολής για να συμπληρώσω την απάντηση του συναδέλφου στην ερώτηση του κύριου Φόξ όσον αφορά εισβολή ή πρόσκληση. Η πρόσκληση έγινε στο πλαίσιο της ε, συμφωνίας που διέπει το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Υπάρχει ένα άρθρο σε αυτή τη συμφωνία που καθιστά όλα τα κράτη αλληλέγγυα. Έναν ένα από αυτά είναι σε κίνδυνο και οι υπόλοιποι θεωρούν ότι είναι σε κίνδυνο και οφείλουν να βοηθήσουν το αντίστοιχο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για να συντομεύω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ισχυριστούν οι αρχές του Μπαχρέν ότι εγώ δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, σας λέω μόνο και κατά την άποψή μου δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι έχουν μπει 2.000 ε, στρατιώτες ξένοι. Όχι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ε, για αυτούς ε, εισβολή. Υπάρχει νομική βάση δηλαδή, υπήρξε πρόσκληση. Και δεν έχω απάντηση, κύριε Πρόεδρε, στο ερώτημά σας για την Αλτζαζίρα με το ποιο τρόπο δηλαδή παρουσιάζει το προβλήματα του Μπαχρέν δεν το γνωρίζω. Δεν έχουμε αντιπροσωπεία εκεί και άρα δεν έχουμε σχετικές πληροφορίες. Και για τη θέση του Κατάρ σε σχέση με την Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα, κανονικά δεσμεύεται από τις ίδιες αλλά δεν έστειλε κανέναν. Ενώ συμμετέχει στην επιχείρηση κατά τη Λιβύης. Νομίζω πως ίσως μοιράστηκαν τα καθήκοντα. Οι Σαουδάραβες και τα Εμμυράτα αποφάσισαν να παρέμβουν στον Παχρέν και η το Κατάρ για δικούς του λόγους θέλησε να μπει στην ε, συμμαχία των προθήμων για τη Λιβύη. Η κυρία Μπράτνα, θα πρέπει να επανέλθω στα σχόλια του κυρίου ε, Κούπερ. Ε, με έχουν ανακουφίσει λίγο αυτά που είπε ο κύριος Μιγκαρέλη. Αυτά που είπατε εσείς ότι είναι ένα ειρηνικό μέρος το Μπαχρέιν ε, και την Ισία ε, ειρηνικό μέρος ε, θα ήταν αρχές Ιανουαρίου. Τι θα πει ειρηνικό μέρος όταν προσπαθεί ο κόσμος να αλλάξει την πολιτική κατάσταση εκεί. Και τι συμβαίνουν ατυχήματα. Έχουν εισβάλει ε, στρατεύματα της Σαουδικής Αραβίας. Δεν είναι ότι έγινε ένα δυστύχημα εκεί. Περίεργος είναι ο τρόπος που τα παρουσιάζετε τα πράγματα. Δεκάδε νεκροί από τη μια πλευρά και μπορεί να έχουν πεθάνει και δύο αστυνομικοί από την άλλη, στρατεύματα που ε, επελάβουν ε, κατά των πολιτών και λέτε ε, συμβαίνουν και ατυχήματα και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ζητώ συγγνώμη, δεν έρχονται σε εμά γαλλικά στρατεύματα όταν έχουμε μαζικέ διαδηλώσει στη Γερμανία να αρχίζουν να πυροβολούν του γερμανού διαδηλωτέ. Ποια είναι τα μέτρα και τα σταθμά που χρησιμοποιείτε. Με τρομάζουν πάρα πολύ αυτά που λέτε. Ε, Ο Βίλι Μέγερ, ευχαριστώ. Κοιτάξτε κύριε Κούπερ, ε, παρεμβάσεις σαν αυτές που κάνατε εδώ είναι αυτές που μας στερούν κάθε αξιοπιστία στον αραβικό κόσμο. Καμία αξιοπιστία δεν έχουμε. Εγώ επιστρέφω από την Αίγυπτο. Είχαμε ακρίβεια πυράβλου κρούς στην καταδίκη του καθεστώτος του ε, Καντάφη, ενώ με τη Σαουδική Αραβία και το Μαγχρέιν δεν κάνουμε τίποτα και αυτό μας καταδικάζει στα μάτια των Αράβων. Εσείς διατηρείτε ίσες αποστάσεις, ε, ε, ισόρροπες και δεν χαρακτηρίσατε ούτε το καθεστώς του Μπαχρέινου ούτε της ε, Σαουδικής Αραβίας. Γλιστρήσατε με τη δικαιολογία. Μα είναι αδικαιολόγητα αυτά που συμβαίνουν. Και το καθεστώς, το φεουδαρχικό της Σαουδικής Αραβίας. Φεουδαρχικό, αντιδημοκρατικό, δικτατορικό και το ε, καθεστώς του Μπαχρέιν. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Είμαστε πολύ ακριβείς, σας επαναλαμβάνω, ακρίβεια πυράβλου κρούζ είχαμε για τον Καντάφη όταν χαρακτηρίσαμε το καθεστώς του. Το ίδια να ισχύουν και για τον Παχρέν και για τη Σαουδική Αραβία. Αυτό που μα λέτε μας αφοπλίζουν τελείως. Α, ότι νεκροί λέτε υπάρχουν κατέρωθαν. Όχι. Δεν είναι έτσι η πραγματική κατάσταση, πιστεύω εγώ. Η πραγματική κατάσταση είναι ότι σήμερα στη Γενέβη η υπατιαρμοστία του ΟΗΕ είπε ότι είναι 50 ή ή αγνοούμενοι. Επιτέθηκαν σε νοσοκομείο. Συνέλαβαν γιατρούς. Γιατρούς συνέλαβαν. Ε, δεν μπορεί κανείς να τηρεί στις αποστάσεις. Θα πρέπει να πούμε στο ε, Μπαχρέν και στο καθεστώς ότι ως εδώ φτάνει πια και να φύγει η Σαουδική Αραβία και να εκδημοκρατιστεί. Και να σταματήσει αυτή η φεουδαρχία. Και η γυναίκα στη Σαουδική Αραβία να ε, θεωρείται άνθρωπος. Αλλιώς δεν είμαστε αξιόπιστοι. Εγώ επιμένω. Δεν σας λέω ότι θα πρέπει να μπουκάρουμε στη Σαουδική Αραβία, ούτε στο Μπαγκρέιν, ούτε συμφωνώ με την επέμβαση στη Λιβύη. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να δράσουμε. Και είπα ότι εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει στάση στεναρή δραστήρια καταδικάζοντας αυτά τα δύο καθεστώτα που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε με το διεθνές δίκαιο. Ε, Κοιτάξτε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, πολύ ζωντανή και νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Είναι λοιπόν, φαντάζομαι, εφικτό να επανέλθει η τάξη, το δίκαιο ε, και κάπως να προστατευτούν οι άμαχοι στη Λιβύη. Αλλά ίσως ε, στον κόλπο αυτά είναι πιο δύσκολο για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Και θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση προς τον κύριο Κούπερ. Ε, δεν ξέρω αν επίτηδες ε, ή κατά λάθο ε, δεν απαντήσατε σε αυτά που σας είπα σχετικά με φήμες που έρχονται από το Ιράν σχετικά με τον Μπαχρέιν ως μια χώρα που έχει δικά συμφέροντα το Ιράν. Εσείς μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε τον Μπαχρέιν, θα το προστατεύσετε με κάθε τίμημα για να ισχύει το διεθνές δίκαιο. Γιατί άκουσα κάτι φήμες ότι το Ιράν προσπαθεί ε, να γίνει ε, πολύ πιο επιθετικό και να ε, εφαρμόσει την πράξη τις αλυτρωτικές του απόψεις. Ναι. Θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον Γκρεγουάρ Τερή τώρα που είναι στην αίθουσα και εκπροσωπεί τη διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Νίμπλερ προηγουμένως μας είπε ότι ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κύριος Ναμπίλ Ραζάμπ του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν είχε ε, ληφθεί και κρατείται. Μπορείτε να μας ενημερώσετε παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να επιβεβαίωσω ότι ο κύριος Ναμπίλ Ραζάπ ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του Κέντρου Μπαχρέν για ανθρώπινα δικαιώματα ε, συνελήφθη την Κυριακή και ήταν και τακτικός συνομιλητής μας, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη ότι πέστη ε, βασανιστήρια και σωματικά και ψυχολογικά με απειλή βιασμού και είναι πραγματικά ε, μέθοδος ε, ε, που ακολουθούν κάποιοι για να συνθλίψουν αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαφανίζονται και γιατροί και αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσπαθούν να τους κάνουν να σπάσουν εντός εισαγωγικών και φοβούνται οι πολίτες να πάνε στο γιατρό μη τυχόν και τους συλλάβουν. Και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο ε, και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ειδικά για τον Παχρέιν, ανησυχούμε λίγο. Ως προς τη διατύπωση ε, που θα ήθελαν ε, οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν καταδικάζουν την απώλεια ζώων αλλά εκφράζουν τη λύπη τους για την απώλεια ζώων στο Συμβούλιο. Αυτό υπολείπεται ε, της διατύπωσης που θα επιθυμούσαν και οι διαδηλωτές και οι ανεξάρτητοι ε, εκπρόσωποι ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να το διαρευνήσουμε και θα σας αναφέρουμε στη συνέχεια. Μα... είναι προς το συμφέρον τους η επαναφορά της τάξης του δικαίου. Ο κύριος Μιγκαρέλη, όχι, μισό λεπτό, ο κύριος Κούπερ θα μιλήσει πρώτα. Ε, κοιτάξτε, δεν ε, κατάλαβα και δεν θυμάμαι καλά τα ονόματα όλων, αλλά θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν και να λειτουργούν κανονικά. Όταν είπα ότι υπάρχουν ε, φήμες και από τις δύο πλευρές για το τι ακριβώς συνέβη, ότι τα νοσοκομεία είναι ένα από τα θέματα όπου δίστανται οι απόψεις. Ε, πρέπει πράγματι να αναζητήσουμε την αλήθεια. Δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού. Εκείνο όμως που δεν είναι αλήθεια είναι ότι οι ε, δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ε, ενεπλάκησαν στις διαδηλώσεις. Όχι, δεν συνέβη αυτό. μπήκαν στο Μπαχρέν μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης του Μπαχρέν. Και είναι αλήθεια ότι ε, είχαμε θανάτους και στις δύο πλευρές, βία που ασκήθηκε εναντί και των δύο πλευρών. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα ονόματα, αλλά συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, στο πίσω μέρος της ε, αίθουσας σχετικά με τον άνθρωπο που συνελήφθη την Κυριακή. Απαράδεκτα βέβαια αυτό που συνέβη. Και νομίζω ότι φοβάμαι ότι ξέχασα την ερώτηση του κυρίου Τάνοκ, γιατί ξέρετε, φοβάμαι ότι την ξέχασα γιατί δεν ξέρω και την απάντηση. Πάντως, ε, στο τέλος, αυτό που ελέγχθη σχετικά με την ε, δέσμευση για την κυριαρχία του Μπαχρέν ως ανεξάρτητου κράτος, προφανώς και ισχύει αυτό, Υπήρξαν βέβαια κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια από την κυβέρνηση του Ιράν, από κάποιους ε, μέσα στην κυβέρνηση του Ιράν. Νομίζω ο εκπρόσωπος τύπου κάτι είπε αυτός για τον Μπαχρέν, ότι θα πρέπει ε, να επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώ του που ήταν η 13η επαρχία του Ιράν. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ε, κανείς να το λάβει αυτό το σχόλιο τόσο σοβαρά υπόψη του επανέρχομαι στο βασικό ερώτημα ότι πράγματι εδώ πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί και πρέπει να λυθεί και θα λυθεί μόνο εάν οι δύο πλευρές συζητήσουν στις προτάσεις που κατέθεσε ο διάδοχος. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μιγκαρέλη, έχω ακόμα έναν εγγεγραμμένο μιλητή, τον κύριο Έλμαρ Μπροκ. Παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Μιγαρέλη να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω ερώτηση για τον Μπαχρέιν εγώ, αλλά για κάτι που βρίσκεται κοντά. Σήμερα το απόγευμα ακούσαμε εκτενέστατη αναφορά για την κατάσταση στην Ιεμένη, όπου πιστεύω συστηματικά εκπρόσωποι του Προέδρου πυροβολούν στο κεφάλι συνειδητά ε, μέχρι ε, νέα παιδιά 13 ετών είναι στα νοσοκομεία από ελεύθερους σκοπευτές, είναι σε βαριά κατάσταση. Είναι συστηματική εγκληματική δράση κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Έχουν προθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εξωτερική Δράση ε, να ε, προχωρήσουν να αναλάβουν κάποια δράση, γιατί δεν βρίσκω διαφορά ανάμεσα στι εγκληματικέ ενέργειε και στι δράσει τη κυβέρνηση Εμένη. Άλλο ένα και ε, η κυρία Μάντνερ. Ο κύριο Μπρόκ σωστά είπε για την ΕΜΕΝΗ. 50, 15 συγγνώμη, εκατομμύρια δίνουμε στην ΕΜΕΝΗ από το μέσο σταθερότητα. Πού πάνε αυτά τα χρήματα, γιατί πηγαίνουν στην κυβέρνηση. Ο κύριο Μεγκαρέλη, ευχαριστώ. Για την Ιεμένη έχει δίκιο ο κύριο Μπροκ. Στη χώρα αυτή, εδώ και εβδομάδε τώρα, είναι δεκάδε νεκροί. Επίση. πού οφείλονται οι δυσκολίε, Μία μειονότητα έχει σφετεριστεί τον εθνικό πλούτο. Η φτώχεια είναι πολύ μεγάλη και ε, ο πρόεδρος Σαλέ είναι ανίκανος να αρχίσει διάλογο με το λαό του. Λοιπόν, χτες είχαμε νέες εξελίξεις. Τρεις στρατηγοί μεταξύ των πιο σημαντικών της χώρας άλλαξαν στρατόπεδο και πήγαν με τους διαδηλωτές. Υπάρχουν επίσης και κάποιοι φύλαρχοι που πέρασαν ε, με τους, στους αντιφρονούντες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο πρόεδρος Σαλέχ απέλησε την κυβέρνηση και πολλοί ε, πολιτικοί του σύμμαχοι σήμερα έχουν αποστατήσει και είναι με την αντιπολίτευση τα πράγματα επιταχύνονται. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να διατηρηθεί για πολύ καιρό η κατάσταση. Έτσι δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να σταθεί στο θόκο του ο πρόεδρος. Ακριβώς επειδή έχει φύγει ένα μέρος του στρατού, ένα μέρος των φιλάρχων και ένα μέρος των πολιτικών του συμμάχων ε, παραδοσιακά έχουν αποστασιοποιηθεί και ε, ε, είναι πολλοί διαδηλωτέ και διαμαρτυρία. Στο βορρά είναι η μειονότητα ούτη που εδώ και αρκετό καιρό έχουν αντάρτικο κανονικό. Ε, επίσης αποσχιστικέ τάσει στο νότο και η νεολαία που εκφράζει τη δυσφορία της και την απόγνωσή της με πολλούς τρόπους και επιπλέον και στη γενιαμένη και αυτό υπάρχει, δεν είναι η αιτία του προβλήματος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θύλακες οργανώσεων ε, τρομοκρατικών. Δεν ελέγχεται το σύνολο της επικράτειας. Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική στην Ιεμένη και κινδυνεύει να επιδεινωθεί η ταχύτητα τις επόμενες ημέρες. Απέναντι σε αυτό θα μου πείτε τι κάναμε. Ε, όπως συχνά δηλώσεις και συμπεράσματα διαφόρων συνεδριάσεων. Υπήρξαν ε, επανειλημμένα δηλώσεις της υπάτης εκπροσώπου για να καταγγείλει τις βιοπραγίες κατά των διαδηλωτών, επανειλημμένα καλούσαμε ε, σε εθνικό διάλογο. Εχθές μόλις ε, μια συνεδρία του ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών με συμπεράσματα που καταδικάζουν την καταστολή και ζητούν διάλογο και ιδιαίτερα η απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Πρόεδρων μας καλεί να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας απέναντι στην Ιεμένη. Ε, ποια πολιτική μας. Από τη μια έχουμε συμφωνία συνεργασίας που εφαρμόζουμε τακτικά και ένα πρόγραμμα βοήθειας. Το πρόγραμμα βοήθειας και απαντώ στην κυρία Μπραντνερ εδώ ουσιαστικά είναι ε, προς όφελος του πληθυσμού άμεσα. Υπήρξε βέβαια ένα σχέδιο αναθεώρησης του τομέα ασφαλείας, αλλά να είστε βεβαία ότι θα το μελετήσουμε πάρα πολύ σχολαστικά. Εμείς τι κάναμε, βοήθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, συνεδρίασαν δύο φορές οι φίλοι της Ιεμένης, μια φορά πέρυσι το Φλεβάρι στη, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη το, πέρυσι το Σεπτέμβριο ε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για καταπολέμηση τρομοκρατίας ήταν πάντα ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της διεθνούς κοινότητας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε σχέδια για την αναθεώρηση και μεταρρύθμιση της ασφάλειας. Να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε σχολαστική και αν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία για την ενδεχόμενη χρήση ε, της βοήθειας της Ένωσης τα καταστολή θα τη διακόψουμε. Για να ολοκληρώσω Πρόεδρε για τον Μπαχρέιν νομίζω αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε μάλλον είναι να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, να ενημερωνόμαστε, γιατί όταν δεν έχουμε επιτόπου αντιπροσωπεία δεν είναι πάντα εύκολο και πριν λαμβάνουμε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται, να αποφεύγουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά, γιατί είναι μόνιμος κίνδυνος αυτό και ε, να μην βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι κυβέρνηση και διαδηλωτές και να δούμε αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που θα οριστεί να παίξει ένα διευκολυντικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Γιατί αν θέλουμε να υπάρχει πραγματικό εθνικό διάλογο, χρειάζεται υποστήριξη ε, έξωθεν. Εάν το επιθυμούν οι ε, πολίτε του Μπαχρέν, γιατί θα πρέπει να μα το ζητήσουν. Και πάλι μέσω κάποιων προσωπικότητων ή κάποιων αντίστοιχων κατάλληλων μηχανισμών μπορούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση και την έναρξη διαλόγου. Bien. Je, je vous remercie. La, la... Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος συνεδρίασης. À quelle heure Ah oui, réunion du bureau élargi à 18h30. 6.30 ώρα διευρυμένο προεδρείο.